Καλησπέρα συνάδελφοι. Σας ζητώ να κάνετε δεκτή την μερίσια διάταξη. Δεν έχω ανακοινώσεις να κάνω. Για τους τριγωνικούς διαλόγους, ο πρώτος πολιτικός για την οδηγία κατά της έκπληξης βρώμικου χρήματος Μητρώα ναι, σε επιχειρηματικές και μειοντότητες ε, where ε, we ε, συνεργασία με FIU για, την, για τους ορισμούς των, των μορφών διαφάνειας. Ο επόμενος τριγωνικός διάλογος θα γίνει στο Στρασβούργο Το θέμα μας σήμερα είναι το PFD2, D2 PSD2 λοιπόν έχει προηγηθεί η δημόσια διαβούλευση Νομίζω ότι είναι έγκαιρη η συζήτηση αυτή γίνεται σε έφετο χρόνο για τα συστήματα πληρωμών θα δώσω το λόγο καταρχάς στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή Μετά θα ακούσουμε και τον βοηθό Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο κ. Ένρια από το EBA έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς ολοκληρώσαμε την προσπάθειά μας, λέει ο κύριος Ένδρια, τον προηγούμενο μήνα. Technical standards on strong uh, customer authentication and secure communication and the very extent και εμείς ε, διαμορφώσαμε μια σειρά από πίνακες οι οποίοι αντικατοπτρίζουν την αξιολόγηση με βάση τις 224 ερωτήσεις, τις περισσότερες που έχουμε πάρει ποτέ μετά από διαβουλεύσεις. Σήμερα θα ήθελα να συγκεντρώσω την προσοχή μου σε τρία βασικά θέματα Καταρχάς ε, ε, τα είχαμε θέσει τον Νοέμβριο. Το πρώτο αφορά τη λεγόμενη τεχνολογική ουδετερότητα, τις εξαιρέσεις ε, από τα επίπεδα ασφαλείας, δημόσια δίκτυα μεταφορών, όπως επίσης και ανάλυση κινδύνου και πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε στα πλαίσια των επιπέδων ΆΙΖΟ, αλλά μετά από τις ανησυχίες οι οποίες έχουν εκφραστεί, ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να βρεθεί μια διαφορετική ισορροπία στον τομέα της καινοτομίας και στον τομέα της διευκόλυνσης και σταθεροποίησης ενός επίπεδου των αγορών. Γνώση λοιπόν, κατοχή στοιχείων και ανείχνευση είναι τα στοιχεία τα οποία θα έλεγα αντιπροσωπεύουν και το ISO 27001. Το πεδίο εφαρμογής ε, ε, είναι κάτι το οποίο καλύπτει συγκεκριμένες βέβαια περιπτώσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένες δυνατότητες εξαίρεσης αλλά έχουμε να κάνουμε για τις ε, αναλύσεις κινδύνου συναλλαγών πλήρη έλλειψη ε, εξαιρέσεων σε σχέση με τις προτάσεις που είχαν γίνει στο έγγραφο διαβούλευσης. Τώρα τα δημόσια δίκτυα μεταφορών και οι αυτοκινητιστική σταθμοί έχουν υπάρξει κάποιες εξαιρέσεις ιδιαίτερα για τους σταθμούς οι οποίοι λειτουργούν πλήρως ηλεκτρονικά θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται το γεγονός ότι οι εξαιρέσει θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν συγκεκριμένους λειτουργικούς λόγους αποφυγής αναμονής υπερβολικής και πιθανών ατυχημάτων στα σημεία ελέγχου. Είχαν πει ορισμένοι ότι το EBA, e η Τραπεζική Αρχή, δεν προέβλεπε αρκετό χώρο για εξαιρέσεις που βασίζονται σε αξιολογήσεις κινδύνου, ιδιαίτερα σε επίπεδο, νομοθετικό επίπεδο 1. Η βασική αρχή, η οποία περιλαμβάνεται στο PSD2, απαιτεί την τραπεζική αρχή να καθορίσει κάποιες, είναι αλήθεια, εξαιρέσεις. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι ε, η πρόταση που γίνεται από ορισμένου εμπλεκομένους στο RTS ε, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην στρέβλωση των κανόνων. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε ότι και η δική σας άποψη σε σχέση με τις εξαιρέσεις που βασίζονται σε ανάλυση κινδύνου συναλλαγών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να καθοριστεί σωστότερα με συγκεκριμένα κριτήρια έχουμε κάποιες δυνατότητες εξαιρέσεων για πληρωμές μέχρι 500 ευρώ και που συνδέονται με ποσοστά απάτης τα οποία καθορίζονται στην πρόταση για το RTS. Βέβαια, τα δεδομένα για απάτες μερικές φορές δεν, τα στοιχεία, επαναλαμβάνω, τα οποία έχουμε δεν είναι πλήρως αντιπροσωπευτικά για τη συγκεκριμένου τύπου εξαιρέσεις. Τώρα για τα ανώτατα επίπεδα εμείς ε, κάνουμε μία πρόταση από τα 10 ευρώ. Ε, θέλουμε εμείς να βελτιώσουμε την ασφάλεια και πιστεύουμε ότι τα θέματα ασφάλειας δημιουργούν και εμπιστοσύνη στις καινοτόμες μορφές ε, πληρωμής. Και αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται εις βάρος των βασικών στόχων του PSD2 όπως της αύξησης της εμπιστοσύνης του καταναλωτή. Εμεί αποφασίσαμε λοιπόν να περάσουμε την εξαίρεση από τα 10 στα 30 ευρώ και δεν φτάσαμε στα 50 ευρώ, κάτι το οποίο ισχύει σήμερα για τις λεγόμενες εισαγωγικά ανέπαφες συναλλαγές between account hmm. Υπάρχει όμως θέμα με τη συλλογή πληροφοριών και την πρόσβαση στους λογαριασμούς πληρωμών. Έχοντας έρθει σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ερμηνεία της συγκεκριμένης οδηγίας, είδαμε ότι η μεταβατική περίοδο για το PSD2 έχει τερματιστεί και το PSD2 δεν αναφέρεται σε αυτό το οποίο ονομάζουμε screen scraping στα αγγλικά. service providers. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει οι εμπλεκόμενοι σε μία συναλλαγή να μην χρησιμοποιούν την πρόσβαση ε, και την σόρευση στοιχείων για άλλους λόγους πέραν αυτών που προβλέπονται από τον κανονισμό για την συγκεκριμένη πληρωμή της Το άρθρο 115 του PS2 προβλέπει ότι οι παροχείς αυτοί έχουν το δικαίωμα να συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς πληρωμών όπως το κάνουν και σήμερα για μία μεταβατική περίοδο περιμένοντας την ημερομηνία εφαρμογής του RTS. Ο μοναδικός νομικά σωστός δρόμος τον οποίο εμείς θεωρούμε ότι έχουμε στην διάθεσή μας σαν EBA απαιτείται να προσφέρετε, απαιτεί να προσφέρετε τουλάχιστον ένα interface και για τις παροχής υπηρεσίες ε, και για αυτούς που εμπλέκονται στη συναλλαγή. Το RTS προβλέπει ότι οι μπορεί να έχουν ένα συγκεκριμένο νέο interface ή να επιτρέπουν ένα προσαρμοσμένο interface για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Όπως και να έχουν τα πράγματα ε, θα πρέπει η ε, ενημέρωση για τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν να είναι εύκολα προσβάσιμη από τους πελάτες. Απαιτείται προσαρμογή σε συγκεκριμένα τεχνικά επίπεδα έτσι ώστε να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο διαθεσιμότητας και επίδοσης το οποίο προσφέρεται στους άμεσους πελάτες τους ε, και ταυτόχρονα να υπάρχουν αντισταθμιστικά εναλλακτικά μέτρα σε περίπτωση μη προγραμματισμένης ε, έλλειψης διαθεσιμότητας. Και θα πρέπει επίσης ε, να υπάρχει άμεση ενημέρωση για το αν τα χρήματα έχουν ε, ήδη καταβληθεί και μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία η συναλλακτική. Απαιτείται λοιπόν να έχουν ε, τις ίδιες πληροφορίες τουλάχιστον από αυτές τις οποίες έχουν στην διάθεσή τους οι καταναλωτές μέχρι τώρα. Θα πρέπει λοιπόν να εναρμονιστεί ακόμα περισσότερο η διαδικασία έτσι ώστε ε, να καλυφθούν οι ανάγκες των χρηστών. Νομίζω ότι στα πλαίσια της εντολής ε, την οποία έχουμε αυτό μπορούσαμε να κάνουμε. Ακούσαμε τα σχόλια που έγιναν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, κάναμε συγκεκριμένες αλλαγές έτσι ώστε να βρούμε μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα σε διαφορετικούς και πολλές φορές αντιθετικούς μεταξύ τους στόχους. Αν τυχόν έχετε ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας. Thank you very much to Andrea I'll give the floor to Pierre Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον Pierre Πετή, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή. Yes. I, I would suggest, if you don't mind, that... Αν δεν σας πειράζει, θα δώσουμε πρώτο λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, καλώς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ελάβαμε το σχέδιο κειμένου των τεχνικών προτύπων πριν από ένα μήνα. Να ευχαριστήσω την Ένωση Τραπεζών για το εξαιρετό έργο της από αυτού και γενικώ θεωρούμε ότι αυτό το σχέδιο κειμένου για το RTS είναι πολύ καλής ποιότητα και επίση συμφωνώ με τον κύριο Ενρία ότι δηλαδή το PSD υπαριθμών 2 κατοχυρώνει αυτούς τους στόχους, γιατί πολλές φορές αυτοί είναι δύσκολο να συγκεραστούν την ασφάλεια, το να είναι βολική ρύθμιση, υποστασία του καταναλωτή, καινοτομία, ανταγωνισμός και νομίζω ότι η Ένωση Τραπεζών ε, έκανε καλή δουλειά σταθμίζοντας όλους αυτούς τους ε, ε, διαφορετικούς στόχους. Σήμερα να μην υψηλούμε σε όλα τα επιμέρους ζητήματα αυτά τα οποία καλύπτει το RDS, αλλά να περιοριστούμε στα ε, εξή δύο. Πρώτον, ασφάλεια και δεύτερον, ε, αυτού του είδους το interface της ε, επικοινωνίας, γιατί είπαμε θέλουμε να υπάρχει η επαλήθευση του πελάτη, επομένως συμφωνούμε με την Ένωση Τραπεζών όσον αφορά αυτόν τον εναλλακτικό μηχανισμό επί τη βάση της ανάλυσης κινδύνων. Και το κάναμε αυτό θεωρώντας ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιος δόκιμος τρόπος επαλήθευσης ε, και αυτό να ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θεωρούμε ότι το RTS πρέπει να έχει αυτή την ρήτρα αναθεώρησης και να υπάρχει κάποια βραχυπρόθεσμη ε, αξιολόγηση όσον αφορά τους μηχανισμούς της επαλήθευσης. Συγκεκριμένα 18 μήνες μετά την εφαρμογή του RTS. Και μετά τους 18 ε, αυτούς μήνες να έχουμε στατιστικά στοιχεία για περιπτώσεις απάτης και κάποια καλύτερα εργαλεία για να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τον κίνδυνο απάτης περί της πληρωμές. Τώρα όσον αφορά το δεύτερο θέμα, δηλαδή ε, αυτού του είδους το interface επικοινωνίας, Βεβαίω. Και δεχόμαστε ότι προσπάθησε να σταθμίσει η EBA τα συμφέροντα των εμπλεκομένων και των τραπεζών, οπότε και συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου. Ότι δηλαδή θα πρέπει να προσπαθήσουμε με το RTS ή με την ερμηνεία του RTS να μην υπονομεύσουμε τους στόχους του PSD2, ότι δηλαδή θα πρέπει να βοηθήσουμε ανταγωνισμό αλλά και καινοτομία. Το σχεδόν κειμένο για το RTS της Ένωσης Τραπεζών η επιβάλληση στι τραπέζε κάποιε υποχρεώσει όσον αφορά την ποιότητα των παρεχωμένων υπηρεσιών. Και με αυτά τα μέτρα όμως θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένα, ούτως ώστε να υπάρχει κάποιο είδου ε, διαρθρωτική αντιστάθμιση για τους ε, παρόχους, τους τρίτους. Και άρα θα πρέπει να γίνει ένα παραπάνω, ούτως ώστε να έχουμε κάποιου είδους plan ε, B, ούτως ώστε οι τράπεζες να μπορούν να προσφέρουν κάποιες εγγυήσεις οι τράπεζες στις ε, επιχειρήσεις. TPP. Τα TPP να είναι βιώσιμα, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει αρκετή ευελιξία για τις τράπεζες. Οπότε κατά αυτόν τον τρόπο νομίζουμε ότι θα βρεθεί μια λύση που θα είναι αποδεκτή από όλες τις πλευρές θα βεβαίω καλή πίστη από όλους. Αλλά θεωρούμε ότι θα τα καταφέρουμε και στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος του κανονισμού της CBA. Ευχαριστώ. Ευχα... Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Γιώργος Και τώρα. Και ε, τώρα έχει το λόγο, κύριε Πετή. Και εγώ με τη σειρά μου να αρχίσω με συγχαρητήρια προς την Ένωση Τραπεζών για όσα έχει κάνει μέχρι τώρα συμπεριλαμβανομένου και του τι έκανε για να διασκεδάσει τις ανησυχίες της αγοράς. Όσον αφορά την πρώτη εκδοχή του κειμένου και επομένως θα πρέπει να υπάρχει ικανή διαφάνεια. Επομένως βρέθηκαν εύστοχες λύσεις σχεδόν για όλα τα θέματα που ασχολούσαν την αγορά και πρόκειται να τις διαβουλεύσει ακόμα. Εκκρεμεί όμω κάτι. Και γι' αυτό να σας πω την απόψη μου. Η πρόσβαση του TPP στους λογαριασμούς των πληρώμων. Σε αυτή την ε, φάση της νομοπαρασκευακής διαδικασίας έχουμε τρεις μεταβλητές. Πρώτα-πρώτα, το τι ανησυχεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και από ό,τι αντιλαμβανόμεθα, αυτό το οποίο σας ανησυχεί είναι το ότι επιθυμείτε το TPP να συνεχιστεί και στο μέλλον. Να συνεχιστεί όσον αφορά το τι γίνεται σήμερα, πώς λειτουργεί σήμερα για την πρόσβαση σε δεδομένα, σε πληροφορίες, όσον αφορά τον λογαριασμό του πελάτη, αλλά και την επιλογή δεδομένων και πληροφοριών ούτω ώστε ο έμπορος να μπορεί να λάβει την επιβεβαίωση του ότι ε, άρχισε η διαδικασία καταβολής του τιμήματος και θα ολοκληρωθεί. Είναι και θέμα ανταγωνισμού όσον αφορά την αγορά λιανικών πληρωμών και αντιλαμβανόμεθα ότι αυτή η λειτουργία θα πρέπει να συνεχιστεί. βεβαίω δυνάμει των όσων επιτάσσει το PSD2 και το ότι τα TPP ή TPP τέλο πάντων να υφίστανται κάποια υποπτία, να είναι εγκεκριμένα και να μπορούν να επισημανθούν πρώτα στοιχεία του οπλευρά των τραπεζών. Επίση, αφού ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, θεωρήσαμε ότι είναι πάρα πολύ θετικό το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή α, πρόκειται να λάβει υπόψη αυτά τα οποία επιζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε κάποια θέματα, να δούμε εντελεχέστερα το θέμα, να δούμε υπό ποιε προποθέσει η πρόσβαση πρόκειται να ε, διατηρηθεί ως ε, εναλλακτική λύση κλπ. κλπ. Τώρα και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Ως και Τράπεζα θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες τραπεζών και των ε, TPP. Και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κοινωνικών Πληρωμών να ξεκαθαριστεί το τι πρακτικές λειτουργίες πρέπει να ρυθμιστούν τόσο ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη αγορά για τις ε, υπηρεσίες πληρωμών στην Ευρώπη. Χρειάζεται ολοκληρωμένη αγορά, ούτως ώστε σε αυτή την αγορά να μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμό μεταξύ των TPP και σε αυτή την αγορά οι έμποροι να μπορούν να χρησιμοποιήσουν μία ή δύο TPP ούτως ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στους ε, λογαριασμούς για τις πληρωμές όσο όλη την Ευρώπη. Λέμε για 4.000 ε, interfaces. Τόσες τράπεζες περίπου υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, εάν η λύση είναι αυτή που τώρα μελετάτε δηλαδή να συνεχιστεί αυτή η δυνατότητα πρόσβασης τότε έτσι θα ξεκαθαριστεί το νομικό πλαίσιο στο οποίο κινούνται οι TPP. Όμως, το θέμα είναι πώς θα βρεθεί ένας τρόπος επικοινωνίας μεταξύ TPP και τραπεζών για όλα τα πρακτικά ζητήματα. Εμείς πάντως πιστεύουμε ότι τελικά θα βρεθεί μια δόκιμη λύση. Άρα συνεχίζουμε να θέλουμε να υπάρχουν αυτές οι κεραυνοβόλες, οι άμεσες στιγμές, πληρωμές και τέτοια λύση να υιοθετηθεί και αυτοί που έχουν παρακολουθήσει τις εξελίξεις γνωρίζουν το πώς ε, εμείς είμαστε υπέρ μιας τέτοιας εξέλιξης όπως γνωρίζετε αυτού του είδους οι στιγμίες ε, πληρωμές θα καλυφθούν από το σύστημα πρόσβασης το οποίο σήμερα συζητούμε. Θα λυθεί το θέμα. Και αυτό θα ρυθμιστεί πριν εφαρμοστεί το RTS το οποίο θα συμβεί κάποια στιγμή το 2019. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Γκολτιέρη για αυτά τα οποία μας είπατε και να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση Τραπεζών διότι έλαβε υπόψη αυτά τα οποία μας απασχολούν. πάρα πολύ ικανοποιητικέ οι προτάσει σας. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και γι' αυτό δίνουμε την σκητάλη στον Φέρμπερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σα ευχαριστήσω και εγώ που έχουν ληφθεί υπόψη κάποιες από τις παρατηρήσεις που κάναμε τότε με τον εισηγητή τον κύριο Ταγιάννη. Ειδικά η τελευταία παρατήρηση με έκανε να χαμογελάσω. Μήπως είμαστε σε θέση με την νομοθεσία μας να ακολουθήσουμε την ταχύτητα ε, με την οποία εξελίσσονται οι εφαρμογές και τα κινητά τηλέφωνα. Λέτε πάντα αυτό στο περιθώριο όσον αφορά τον τριμερή διάλογο. Ε, είναι σαφές όσον αφορά την ε, δεύτερη οδηγία για τις υπηρεσίες ε, πληρωμών. Από τη μία θα πρέπει να είμαστε με το πλευρό των επιχειρήσεων, από την άλλη θα πρέπει να έχουμε και προστασία το καταναλωτή και όσο γίνεται πιο εύκολο τρόπο πληρωμών. Έχουμε λοιπόν εδώ το πρώτο επίπεδο και πρέπει να φροντίσουμε να μπορούν να γίνονται με ασφαλή τρόπο οι συναλλαγές. Η δεύτερη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών ε, επίσης ε, πρέπει να εφαρμοστεί με τρόπο ουδέτερο ως προς την τεχνολογία και τα πρότυπα. Ε, δίδεται εδώ ένα πρότυπο ίσο, το οποίο όμως δεν διασφαλίζει την ουδετερότητα. Επίσης, τα σημεία η αιτιολογική σκέψη 93 αναφέρεται στην πρόσβαση ε, στους λογαριασμούς των πελατών, αλλά αυτό προϋποθέτει όλες οι άλλες προϋποθέσεις να πληρούνται. Δηλαδή, ο τρίτος πάροχος υπηρεσιών ε, πληρωμών θα πρέπει σαφώς να ταυτοποιείται. Θα πρέπει δηλαδή να είναι σαφές εάν ε, παρεμβαίνω εγώ ή κάποιος τρίτος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών. Επίσης, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω μάλλον να κάνω μια παρατήρηση προς την Κομισιόν όσον αφορά την εφαρμογή ε, τη, των εκτελεστικών ε, μέτρων. Μακροπρόθεσμα, νομίζω ότι ε, έχουμε ένα μοντέλο που ε, υπόσχεται πολύ περισσότερα, ε, που πάλι θα έχουμε screen scraping ή να έχουμε συνδυασμό των συστημάτων αυτών. Το πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά θα πρέπει να το εξετάσουμε ήδη τώρα. Δεν μπορούμε να δίνουμε στον ε, πελάτη πλήρη πρόσβαση στον λογαριασμό, αλλά περιορισμένη πρόσβαση στον ε, πάροχο ε, των υπηρεσιών πληρωμών. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να έχουμε ισορροπημένη προσέγγιση και θα παρακαλούσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει οι υπηρεσίες έναρξης πληρωμών και οι υπηρεσίες τραπεζικών λογαριασμών να είναι καλά ισορροπημένε μεταξύ του και να έχουμε ίσες συνθήκες ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το δεύτερο θέμα το οποίο επίσης θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών έχει υιοθετήσει πολλέ από τι αιτιολογικές μας σκέψεις, έχει ε, υιοθετήσει τα κατόφλια που θέλαμε εμείς, ε, καθώ ε, και το θέματα ταυτοποίηση των πελατών. Έχουμε όμως πρόβλημα όσον αφορά τις απάτες εξαιρούνται από το σύστημα ταυτοποίησης των πελατών οι συναλλαγές μέχρι 500 ευρώ. Αυτό σίγουρα είναι καλό για τον ιδιώτη καταναλωτή και σημαίνει ότι φροντίζουμε και για προστασία των καταναλωτών. Από την άλλη όμως γνωρίζουμε ότι κάποια κεντρικά σημεία Εκαθάριση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τραπεζών, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών κλπ. Ε, ε, είναι αρμόδιοι για ε, επαγγελματικά ταξίδια, κάτι που πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά και δεν ταιριάζει σε όλο το πλαίσιο αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε μία ρύθμιση για λύσεις επιχειρήσεων προς επιχειρήσεις, B2B, business to business. Δεν νομίζω ότι κάθε Ευρωπαίος Επίτροπος κάθε μέρα θέλει να δίνει τους κωδικούς των τραπεζικών του λογαριασμών κάθε φορά που πηγαίνει επαγγελματικό ταξίδι. Θα χαιρόμουν λοιπόν πολύ εάν θα μπορούσατε να συμπεριλάβετε και αυτά τα σημεία στην πρότασή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, Κλουβ Δίξον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπα, θα πρέπει και στη συνέχεια να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα ε, των τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ε, να έχουν ε, πρόσβαση στον λογαριασμό του πελάτη μέσω της διαπαφής της τράπεζας στο διαδίκτυο. Η ε, υπάρχουσα εκδοχή των κανονιστικών τεχνικών ε, προτήτων ε, επιτρέπει στην τράπεζα να το αποφασίσει αυτό, αλλά δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τη γνώμη της τράπεζας. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών εντός της εντολής της να βρει ένα καλό τεχνικό μοντέλο. Η αιτιολογική σκέψη 93 λέει ότι ε, οι οδηγίες υπηρεσίες πληρωμών 2 θα πρέπει να είναι συμβατοί με διάφορες τεχνολογικές λύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε ε, εάν ε, μια τράπεζα χρησιμοποιεί ε, ειδική διεπαφή, αυτή να μην βασίζεται σε μοντέλο παράκαμψης, διότι αυτή η τεχνολογία δεν επιτρέπει ε, στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να αναπτύξουν τις δικές, τα δικά τους προϊόντα και να τα προσαρμόσουν σε διάφορα περιβάλλοντα, όπως είναι οι διάφορες εφαρμογές και τα κινητά τηλέφωνα. Επίσης, θα πρέπει να αφαιρεθεί από το κείμενο το πρότυπο ISO 222, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 των κανονιστικών τεχνικών ε, προτύπων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Είναι περίεργο η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να δίνει τεχνικά πρότυπα, ενώ κατά τα άλλα θέλουμε τεχνολογική ουδετερότητα και καινοτομία. Η εισαγωγή του συγκεκριμένου προτύπου σημαίνει ότι η δυνατότητα των τραπεζών να παρέχουν την καλύτερη δυνατή διεπαφή αφαιρείται. Και επίσης ε, αφαιρείται και η δυνατότητα για προσαρμογή των εφαρμογών της τράπεζας στα διάφορα περιβάλλοντα. Το άρθρο 27.4 των κανονιστικών τεχνικών προτύπων ε, λέει ότι ε, διεθνείς οργανισμοί τυποποίησης θα πρέπει να αναπτύξουν πρότυπα για το PIS και AIS. Και πάλι αυτό αντίκειται στην ιδέα της τεχνικής τεχνολογικής ουδετερότητας που διέπει την ε, οδηγία για τις υπηρεσίες πλειομόνη. Είμαι πεπισμένος ότι δεν ε, ε, συμπεριλαμβάνεται στην εντολή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών να δίνει σε τέτοιους οργανισμούς η επίσημη θέση κατά την εκπόνηση διαφόρων προτύπων. Επίσης, θα πρέπει η τεχνική SWIFT να μπορεί να επιβάλλεται στις ε, υπηρεσίες έναρξης ε, πληρωμών, ε, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα ρίξει έξω από την αγορά λόγω του υψηλού κόστου σε διάφορους οικονομικούς παράγοντες και αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ιντβελτ. Θα είμαι σύντομη. Δεν θα μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες. Θα ήθελα να αντιδράσω λίγο σε αυτά τα οποία είπε περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο νομοθετούμε. Ότι δεν είναι κατάλληλος ο τρόπος αυτό σε σχέση με τις ανάγκες. Αναρωτιέμαι λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια που συζητάμε τις τελείες και τα μικρά κόμματα κείμενα τι δυναμικό χάσαμε. Πέρα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου θέματος, το θέμα τίθεται με πολιτικό τρόπο. Αν και για το συγκεκριμένο δεν είμαι απόλυτα σίγουρη για την πρόταση, το θέμα είναι να διασφαλίσουμε την καινοτομία και τον ανταγωνισμό γιατί μέχρι τώρα οι προσπάθειές μας οδηγούν την καινοτομία εκτός Ευρώπης και μετά παραπονούμεθα ότι εξαρτώμεθα από οι Κινέζους και οι Αμερικανούς γίγαντες της τεχνολογίας. Συνεπώς λοιπόν ελπίζω τα μελλοντικά θέματα να αντιμετωπιστούν με καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ. Ίσως να τίθεται σε αμφισβήτηση το ότι η πλήρης απορρίθμιση διασφαλίζει σωστές και εύρυθμες αγορές αλλά εν πάση περιπτώσει είναι επίσημη η πολιτική αυτή. Από την Γκουε όχι, η Ζολή δεν είναι εδώ από τους Πρασίνους, ο Γκίγκολντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, θυμάμαι, ίσως το θυμάται και η Σοφή, ότι όταν διαπραγματευόμεθαν τη ΣΕΤΑ, είχαμε κάνει μια μακρά συζήτηση για τα θέματα διακυβέρνησης της αγοράς και αν δεν καλά, οι λύσεις οι οποίες δόθηκαν για μένα δεν ήταν διόλου μα διόλου ε, ικανοποιητικές. Νομίζω ότι αυτό το οποίο μέχρι τώρα έχουμε κάνει στα πλαίσια της προετοιμασίας είναι η σημασία την οποία έχουν τα interface στα πλαίσια του ERPB. Ένα σώμα δηλαδή το οποίο αντικαθιστά το Συμβούλιο ΣΕΠΑ και το οποίο έχει έδρα την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Υπάρχει μια ιστοσελίδα κεντρική του συγκεκριμένης υπηρεσίας και αν δείτε ε, τον κανονισμό λειτουργίας ε, παίρνει αποφάσεις με πλειοψηφία τριών τετάρτων, κάτι το οποίο σημαίνει ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των ιδίων των τραπεζών. Ε, η γραμματεία παραμένει στο EPC που το οποίο είχαμε κατηγορήσει ότι δεν είναι διαφανές και αντικειμενικό προς όλους τους εμπλεκομένους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχει ισχυρή εκπροσώπηση των ομάδων των καταναλωτών και χρηστών. Και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή δεν είναι καν μέλος. Ε, να μας πει λοιπόν προσκαλείται στις εργασίες του σώματος αυτού. Έχω την αίσθηση ότι το σύνολο της διακυβέρνησης της αγοράς σε σχέση με τις πληρωμές είναι ανεπαρκές και όπως είπε και ο εισηγητής το θέμα είναι να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις αυτές και να μην ασχολούμεθα κατά περίπτωση με το τι συμβαίνει. Έχω την αίσθηση ότι αυτός ο τρόπος διακυβέρνησης είναι ιδιαίτερος περίεργος και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει γιατί αυτή η κομβική ομάδα εργασίας για την εφαρμογή του PSD2 έχει μια γραμματεία η οποία εντάσσεται στο EPC. Και στον κατάλογο των μελών της γραμματείας αυτής υπάρχουν δύο μεγάλες τράπεζες, και ανήκουν σαν μέλη στο EPC και επίσης και ο αντιπρόεδρος της ομάδας αυτής είναι από το EPC. Αυτή η μορφή διακυβέρνησης εμένα μου δημιουργεί μια κάποια δυσφορία. Λοιπόν, γνωρίζουμε ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, γνωρίζουμε ποιος είναι ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας και ψηφίζουμε εμείς τον προϋπολογισμό. Εδώ έχουμε ένα όργανο ανεξάρτητο με πολλούς ρόλους, πολλές αποστολές, αλλά δεν έχουμε το ίδιο επίπεδο ελέγχου και προσπαθούμε εδώ να δούμε τι θα κάνουμε μέσω του EBA, της Τραπεζικής Αρχής, η οποία δεν είναι καν στον κατάλογο των επίσημων των μελών. Συνεπώς λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ, ποιος παίρνει αποφάσεις. Να μας διευκρινίσετε παρακαλώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει αν αυτή η μορφή διακυβέρνησης είναι η διαφανέστερη και η πλέον δημοκρατική στο τομέα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βάλλη δεν είναι παρόν. Όχι. Ξεκινάμε το Catch the Eye. Η κυρία Μπερέσα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να συζητήσουμε το RTS στα πλαίσια της διαδικασίας ελέγχου. Είναι κάτι το σημαντικό το ότι μπορούμε να το επανεξετάσουμε. Έχω την αίσθηση ότι η στάση της EBA, ανεξάρτητα από τη θέση της στην ομάδα εργασίας, είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά ισορροπημένο. Σε πρώτο επίπεδο η βασική ιδέα είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια δυνατότητα ένταξη στην αγορά. Και ανάμεσα στην προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες και στην επιθυμία θα έλεγα των ε, πελατών να χρησιμοποιούν μεθόδους πληρωμής ασφαλής και η διασφάλιση θα έλεγα συγκεκριμένων συνθήκων που προστατεύουν τους καταναλωτές μας κάνουν να σκεφτούμε ακριβώς τους όρους με τους οποίους προτείνονται οι αλλαγές. Κάποιες παρεμβάσεις έχουν σαν στόχο να καλύψουν αν θέλετε αυτούς οι οποίοι εξ των νέων τεχνολογιών ε, επιχειρούν στον συγκεκριμένο τομέα. Η τεχνολογική ουδετερότητα στην ουσία εκλαμβάνεται σαν κάτι αποκλειστικά προς υπηρεσίαν αυτών που είναι ήδη στην αγορά. Το θέμα είναι, θα έχουμε πρόσβαση στα απαραίτητα στοιχεία για τις πραγματικές πληρωμές ή μήπως μέσω απλά των συγκεκριμένων πληρωμών αδειοδοτούμε νέες επιχειρήσεις ή ε, και παλαιότερες να συλλέγουν το σύνολο των πληροφοριών που συνδέονται με τους τραπεζικούς λογαριασμούς πληρωμών. Είναι ένα λοιπόν από τα θέματα τα οποία είχαν τεθεί σε συζήτηση. Είναι κρίμα που δεν υπήρξε μια πραγματική θα έλεγα αντιπαράθεση ανάμεσα σε μεγάλες εταιρείες όπως η Software όπως και κάποιες άλλες περιπτώσεις όπως ε, του τύπου γκάφα που επιτρέπουν στα πλαίσια της τεχνολογικής ουδετερότητας να ενδιαφέρονται από τον έλεγχο των συγκεκριμένων δεδομένων κάτω από όρους και συνθήκες όμως των οποίων το εύρος δεν μπορούμε να προσμετρήσουμε και που διαφεύγουν νομίζω του πνεύματος του νομοθέτη επίπεδου 1 η θέληση του νομοθέτη δεν θα πρέπει να αγνοηθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν η τεχνολογική ουδετερότητα την οποία επιζητούν και οι μεν και οι δε δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να ενισχύεται η θέση αυτών οι οποίοι ήδη είναι ενταγμένοι στις αγορές και δεν θα πρέπει επίσης καθιστώντας εύκολη την κλίδα εισόδου να ευνοήσουμε συγκεκριμένα συμφέροντα. Για το θέμα της ασφάλειας, ευχαριστώ τον κύριο Ανδριά. Ε, εγώ ήμουνα υπέρ των 10 ευρώ, του ορίου ανωτά του 10 ευρώ. Γιατί η ενδιάμεση πληρωμών δεν είναι στην πρώτη γραμμή πολέμησης της τρομοκρατίας, παρόλα αυτά είναι ένα μέσο θα έλεγα ε, σημαντικό που μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ στα τομέα της ασφάλειας. Και όσο περισσότερο ανεβάζουμε το επίπεδο εξαιρέσεων, τόσο θα έλεγα επιτρέπουν να αναπτύσσονται κίνδυνοι οι οποίοι στη συνέχεια θα, για τους οποίους θα υπάρξουν κατηγορίες εις βάρος και των δημοσίων αρχών και των νομοθετικών αρχών όπως ημών των ιδίων. Συνεπώς λοιπόν σε σχέση με τις τεχνολογικές δυνατότητες τις οποίες διαθέχουμε και σε σχέση με τα μέτρα προστασίας του καταναλωτή και της αύξησης της δυνατότητας του καταναλωτή να χρησιμοποιεί τις μέγιστες δυνατές νέες εξελίξεις, πρέπει να πούμε ότι η πρόταση της CBA είναι μια καλή πρόταση και θα βασιστούμε πάνω σε αυτήν για να προσπαθήσουμε να δούμε ποια θα είναι η τελική μας απόφαση. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Δεν έχουν ζητήσει λόγο, οπότε θα σας πει ο υποφαινόμενος δύο λόγια. Βεβαίως, όπως προείπα, θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ πιστικά τα όσα μας είπε ο κύριος Ρέα. Και επίσης να ευχαριστήσουμε την ΔΕΗ για τόσο είπα, διαδόσα αλλά όσον αφορά το πρόβλημα της πρόσβασης στους λογαριασμούς, επ' αυτού θα πρέπει η Ευρωπαϊκή να μας πει τι εννοεί ότι θέλει δηλαδή να επιφέρει κάποιες ε, τροποποιήσεις τόσο ώστε να περιφρουρήσει την σημερινή ε, πρακτική. Δεν θέλουμε να υπονομεύσουμε την ομοθετική ρύθμιση, αλλά βεβαίως και θα πρέπει να συμμορφωθούμε με τους στόχους της νομοθεσίας. Όχι δηλαδή να προστατεύσουμε το επιχειρηματικό μοντέλο μας, αλλά θα πρέπει να υπόψη τις αρχές μας, δηλαδή ισορροπία, ε, ουδετερότητα, ασφάλεια, θεμητέοι όρια ανταγωνισμού και γι' αυτό δεν καταλαβαίνω τι εννοείται αμφισβητώντας αυτό που είπε η EBA δηλαδή αυτό το screen scraping, το οποίο δεν θα επιτρέπεται πλέον δύναμη της ε, νέας νομοθεσίας. Και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι σαφές από το νέο νομοθέτημα. Θα πρέπει να συνεχίσει την ε, λειτουργία αγορά, αλλά δεν θα πρέπει να καταπατούμε αυτή την βασική αρχή που διέπει την νομοθεσία. Οπότε ε, προσωπικά ως μέλος της Επιτροπής θα σας ζητήσω να μας διευκρινίσετε τι εννοείτε ότι θέλετε να τροποποιήσετε αυτό το τελευταίο. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει καμία τροποποίηση. Ευχαριστώ. Thank you, Chairman. Uh, as I said, we... Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Όπως προείπαμε, θεωρούμε ότι το RDS το έχει επεξεργαστεί πάρα πολύ ποιοτικά η Ένωση Τραπεζών και με αυτό το interface επικοινωνίας θεωρούμε ότι θα έχουμε και μπορούμε να έχουμε για τις TPP επιπλέον προστασία. Και έτσι το επιχειρηματικό μοντέλο και η συνέχεια αυτού να εξασφαλιστεί να υπάρχει βιωσιμότητα. Επίσης όσον αφορά την λύση που μελετούμε ε, σημαίνει ότι είτε θα δώσουμε πρόσβαση στις TPP μέσω του interface επικοινωνίας των πελατών και βέβαια μπορούν να υπάρχουν κάποιες προσαρμογές για να έχουμε την ε, σωστή ταυτοποίηση απλώς τραπεζών και TPP και θα εξασφαλίσουμε ότι η TPP θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ή αυτό μπορούμε να κάνουμε επομένω αφενό. Ή από την άλλη μεριά θα μπορούσαν να έχουν τράπεζε ένα ε, ad hoc interface, αυτό το οποίο δεν ορίζεται στο αρτίες, αλλά ε, χρησιμοποιείται από την πλατφόρμα που χρησιμοποιείται τώρα. Επομένως, να έχουμε αυτό το API και επίσης να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τον τρόπο επικοινωνία και να μπορεί να υπάρχει ταυτοποίηση από πλευρά των τραπεζών και φιλτράρισμα των πληροφοριών. Γι' αυτό και είπαμε ότι σκεπτόμαστε το τι θα επιλέξουμε αφού ακούσουμε όλες τις απόψεις εδώ στο Κοινοβούλιο και αφού ακούσουμε όλες τις απόψεις που εκφράζονται στο Συμβούλιο και να δούμε πώς θα γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των επιμέρους απόψεων. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Κεντρική Τράπεζα. Σας ευχαριστώ. Ήθελα να σχολιάσω την παρατήρηση για το RPB. Όπως γνωρίζετε, πρόκειται για έναν φορέα όπου προεδρεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όπου συμμετέχουν διάφοροι παράγοντες, όλοι οι σχετικοί παράγοντες και από την πλευρά προσφοράς και ζήτησης. Ε, συμμετέχουν ε, καταναλωτές, επιχειρήσεις, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τράπεζες, οργανισμοί πληρωμών συμπεριλαμβανομένων των TPP, των τρίτων δηλαδή. <coughs> Εμείς λοιπόν είμαστε πεπισμένοι ότι έτσι διασφαλίζουμε την ε, δίκαιη εκπροσώπηση όλων ε, των συμφερόντων. Όπως είπατε, ε, αυτό το Συμβούλιο, του RPB, έχει δικούς του κανόνες. Όταν δημιουργείται λοιπόν ομάδα εργασίας, όπως για τις υπηρεσίες έναρξης πληρωμών, συνήθως συμπροεδρεύεται από εκπρόσωπο από την πλευρά της ζήτησης ε, και από την άλλη από την πλευρά της προσφοράς. Οι κανόνες και η εντολή της ομάδας αυτής διασφαλίζει να μην διαμορφωθεί καμία λύση από την ίδια την αγορά, διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προεδρεύει, αλλά στόχο έχει να βρίσκει την κατάλληλη λύση. Δεν θα προκύψει καμία λύση από την ομάδα εργασία αυτή εάν δεν αντικατοπτρίζει μια ευρεία συνένεση. Έτσι λοιπόν στο συγκεκριμένο θέμα δεν θα προέλθει λύση από το ERPB που να μην στηρίζεται από όλους τους σημαντικούς παράγοντες στον τομέα αυτών που συμπεριλαμβάνει τράπεζες φυσικά, όχι μόνο τις τράπεζες όμως, αλλά και τους τρίτους οργανισμούς πληρωμών και επίσης προτού να, δώσω, προτού να δώσετε το λόγο στον Αντρέα και ε, το DBA, Είμαστε παρατηρητές στους διάφορους ε, φορείς ε, και όποτε θέλει να συμμετάσχει το TPA στη συζήτηση, η πόρτα είναι ανοιχτή για αυτούς. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τον λόγο ε, στον Τιρκ που συμμετέχει περισσότερο στις τεχνικές εργασίες από ότι εγώ. Θα μπορέσει να σας δώσει καλύτερη εικόνα. Όσον αφορά όμως τις γενικές παρατηρήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση αυτών των προτύπων και για τη διακυβέρνηση. Όσον αφορά λοιπόν το χρονοδιάγραμμα, η εντολή μας είναι όπως δείχνει και η σημερινή συζήτηση, ε, είναι ένα από τα πιο δύσκολα έργα που είχαμε. Είχαμε λοιπόν τον υψηλότερο αριθμό απαντήσεων στη διαβόλευση από ό,τι είχαμε ποτέ. Ε, και έχουμε καθυστερήσει μόλις έναν μήνα. Ε, είμαστε στο 13ο μήνα δηλαδή. νομίζω λοιπόν ότι ήμασταν πολύ πειθαρχημένοι ε, στις εργασίες μας και δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικά επαχθή στη διαδικασία από τη δική μας πλευρά. Όσον αφορά τη διακυβέρνηση, ούτε γνώριζα για την ομάδα. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ε, τι στόχο έχει. Έχουμε τις δικές μας δομές και συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως άλλωστε απαιτείται από μας αλλά συμμετέχουν στην ομάδα εργασία αυτή μόνο δημόσιες αρχέ από ό,τι κατάλαβα. Μετά έχουμε τη δική μα ειδική ομάδα για τι υπηρεσίε πληρωμών. Αυτοί είναι οι φορεί που εκπώνησαν ε, τα πρότυπα αυτά και νομίζω ότι πολύ σωστά έγινε αυτό έτσι. Εάν υπάρχουν ε, άλλες επαφές ε, με τον οικονομικό τομέα, αυτό είναι καλό, αλλά νομίζω ότι καλύτερο είναι να μην συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στις εργασίες αυτές. Έχουμε κανάλια για τις ε, δημόσιες διαβουλεύσεις ε, και νομίζω ότι είμαστε ε, διαφανείς όσον αφορά τις επαφές μας με ιδιωτικούς φορείς. Ντίρκ, θα σου ζητούσα να απαντήσεις σε τεχνική παρατήρηση που έγινε για τη διεπαφή. Αλλά γενικά νομίζω ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη λύση εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Είναι όμως απαραίτητο να βρούμε τρόπους ώστε οποιοδήποτε έχει πρόσβαση σε λογαριασμό πελάτη να πρέπει να ταυτοποιείται και να παρέχονται επαρκή εχέγγυα όσον αφορά την ασφάλεια και να εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή της υπηρεσίας που έχει ζητήσει ο πελάτης. Τα πρότυπά μα λοιπόν, ε, ευθυγραμμισμένα και με την ομοθεσία προσπαθούν να πετύχουν ακριβώ αυτό. Αλλά, Ντίρκ, ε, εάν μπορεί να απαντήσει και στην ερώτηση που έγινε σχετικά με τα 500 ευρώ. Σύντομα σας παρακαλώ, διότι πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. 30 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα. Από θέσεις από εσά ε, ακούσαμε σχετικά με την ε, διαδικασία ανάπτυξης της πολιτικής αυτής. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι προχωράμε σε νέα μοντέλα και πρώτη φορά Έχουμε τις ε, απαιτήσει ασφαλείας στην νομοθεσία. Ε, έχουμε ξεκινήσει λοιπόν μια πολύπλοκη διαδικασία. Έχουμε μάθει πολλά και πολύ ευχαρίστω θα τα εφαρμόσουμε. Εμάς όμως δεν μας εκπλήσει η θέση στην οποία βρισκόμαστε, διότι είναι μεγάλο βήμα η συμπερίληψη στην νομοθεσία των απαιτήσεων περί ασφαλείας. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, όπως είπε και ο Ανδρέα, καθυστερήσαμε ένα μήνα. Είχαμε ε, διαβούλευση, είχαμε και έγγραφο συζήτησης για να είμαστε βέβαιοι ότι καταλαβαίνουμε και εμείς με τον ίδιο τρόπο την οδηγία ε, όπως και οι αγορές. Εάν υπάρχει κάποια ανησυχία, έχει να κάνει με το 18μηνο που προβλέπει η ίδια η οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών. Ε, το 18μηνα δηλαδή μέχρι την θέση σε ισχύ της οδηγίας. Αυτό δεν είναι κάτι που το έχουμε αποφασίσει εμείς. Ε, αυτό έχει θεσπιστεί εντός της οδηγίας. Μπορεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, αλλά νομίζω ότι ε, προς στιγμήν ε, έχουμε, έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες μας εγκαίρως για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε την αγορά. Όσον αφορά αυτό που και νωρίτερα σχετικά με την πρόσβαση στους ε, λογαριασμούς, ε, η τεχνολογική ουδετερότητα ε, ορίζεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Εμείς θέλαμε να φροντίσουμε να μην έχει πιο ευνοϊκή μεταχείριση κάποιος, ε, κάποιος παράγοντας από κάποιον άλλον. Και πιστεύουμε ότι το έχουμε πετύχει αυτό μαζί με τους άλλους 7 μας στόχους. Δηλαδή η τεχνολογική ουδετερότητα είναι ένας από 8 στόχους. Ε, και εσείς παρακαλώ πολύ σύντομα. Να είμαι ειλικρινής, ε, ε, έχω απογοητευτεί πολύ. Δεν απαντήθηκαν οι ερωτήσεις μου, καμία από τις ερωτήσεις μου δεν απαντήθηκαν. Το θέμα διακυβέρνησης ε, δεν είναι ε, θέμα των ε, κανονιστικών τεχνικών προτύπων, RTS. Και επίσης είμαι απογοητευμένος που θεωρήθηκαν σημαντικές ερωτήσεις άλλες από αυτές που έθεσε η διαπραγματευτική ομάδα. Και αν είναι έτσι, να παραιτηθώ από εισηγητής. Δεν έχει νόημα να κάνω τόση δουλειά και να θεωρούνται ξαφνικά ε, ένα σωρό άλλα πράγματα πιο σημαντικά από αυτά που βρίσκονται εντός του πεδίου εφαρμογής των κανονιστικών τεχνικών προτύπων. Και αν αυτό είναι ο τρόπο που χειριζόμαστε τα θέματα εδώ στην Επιτροπή, θα σταματήσω τότε να, τη δουλειά μου, διότι αυτό είναι απαράδεκτο. Ευχαριστώ πολύ. Μάρκους, είναι σαφές, ε, δόθηκε ο λόγος σε όλους, όλοι είχαν τη δυνατότητα να μιλήσουν. Εάν υπάρχουν ε, θέματα που δεν απαντήθηκα, θα ζητήσουμε γραπτώς την ε, απάντηση. Ναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι ε, σήμερα έχουμε την ώρα για την εξέταση των θεμάτων αυτών. Εάν λοιπόν θεωρηθούν ένα σωρό άλλα θέματα πιο σημαντικά, Ε, τι είναι προφανές όμως, ε, λέει ο Πρόεδρος. Ε, λέω ότι η συζήτηση αυτή δείχνει ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις εντός του Κοινοβουλίου και αυτό θα πρέπει να το λάβει υπόψη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαι βέβαιος ότι θα πρέπει να έχουμε και περαιτέρω συζητήσεις πάνω στο θέμα αυτό και εντός του Κοινοβουλίου για να διαμορφωθεί η θέση του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. My uh, Ο Πρόεδρος. Καθίστε παρακαλώ. Μάρκος, please. now... ευχαριστώ. Πάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών πέντε σημείες διαδιατάξεως και ας ευχαριστούμε ένα θερμό κλωσόρι στον κύριο Στράβκο Μάριτς, Υπουργό Οικονομικών της Κροατίας, ο οποίος απεδέχθη την πρόσκλησή μας για να έρθει να μας μιλήσει για το πώς ε, έχει η οικονομική κατάσταση στην χώρα του, τι γίνεται με τις ε, προοπτικές της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι η Κροατία, η χώρα η οποία πιο πρόσφατα ε, προσεχώς στις Ευρωπαϊκές, δηλαδή το 2013, όπως και άλλες, άλλες χώρες. Έλαβε ράπισμα από την χρηματοοικονομική κρίση και η χώρα εκείνη. Στα πλαίσια αυτά δε υπάρχει η μελέτη της κατάστασης. Η κατάσταση τώρα έχει βελτιωθεί. Το έλλειμμα είναι αρκετά κάτω από το 3% του ΑΕΠ και επομένως θα διαπιστωθεί οριστικά τον Μάιο κατά πόσο θα βγείτε από την ε, διαδικασία του ελέγχου των δημοσιονομικών από την Επιτροπή Έχουμε βέβαια τις ε, αναχώρες συγκεκριμένες ε, συστάσεις και για την κατάσταση των τραπεζών. Οπότε πρόκειται για συζήτηση πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα. Έχετε το λόγο. Ο κύριος Μάριτσο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, πρώτα πρώτα επιτρέψτε μου να σας πω το πόσο θετικό θεωρώ το ότι μου δώσατε την ευκαιρία να έρθω και να σας μίλησω και να είμαι ο πρώτος υπουργό των ε, οικονομικών που απευθύνεται στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως ε, προανέφερε ο κύριος Πρόεδρος, θα σας μιλήσω για τις οικονομικές ε, τάσεις και προοπτικές της χώρας μου. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι Είμαι περίφανος που είμαι Κροάτης, αλλά να σας τα πω επόμενος γι' αυτό στα κροατικά. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, για μένα είναι χαρά αλλά και τιμή το να σας μιλώ. Για πρώτη φορά έρχεται εδώ ένας ε, Υπουργός Οικονομικών της ε, Κροατίας να μιλήσουμε για κάποια σημαντικά ζητήματα που αφορούν την οικονομία της ε, Κροατίας, να δούμε και ποιες είναι οι οικονομικές τάσεις για το μέλλον και ακριβώς όπως προείπε ο Πρόεδρος και εμείς όπως και άλλες ε, χώρες περάσαμε ε, πάρα πολύ δύσκολα λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης και της έφεσης ύφεση συγγνώμη που κράτησε έξι χρόνια και μπορούμε πούμε ότι υπήρχε και υπήρξε και σορευτική ε, πτώση του ΑΕΠ μας κατά 12%. Επομένως, σε πολλούς κλάδους της οικονομίας έγινε η κρίση της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας. Ακριβώς γιατί μειώθηκε η οικονομική δραστηριότητα. Οπότε και είδαμε να υπάρχουν πτωτικές τάσεις και στην αγορά απασχόλησης, οπότε και αυξήθηκε η ανεργία. Μειώθηκαν οι απασχολούμενοι, αλλά και υπήρξε επιδείνωση της οικονομικής μας θέσης, ε, ιδίως όσον αφορά τα δημιουργικά. Έχουμε όμως διάφορα προβλήματα, διάφορες ε, προκλήσεις όσον αφορά το δημογραφικό μέτωπο. Νομίζω ότι ξέρετε το ότι αποφασίσαμε ως κυβέρνηση για το ότι τα δημοσιονομικά και τα οικονομικά θα είναι η κορυφαία μας προτεραιότητα. Σας μιλώ τώρα εξ ονόματος των δύο τελευταίων κυβερνήσεων. Βέβαια η προηγούμενη κυβέρνηση κράτησε λιγότερο από ένα χρόνο. Αλλά εν πάση περιπτώσει μπορώ να μιλήσω και για εκείνη την κυβέρνηση γιατί ήμουν και τότε υπουργός οικονομικών. Επομένως και τότε και τώρα είναι κορυφαία προτεραιότητα τα οικονομικά. Το 2016 ήταν καλή χρονιά για την Κροατία. Να σας πω κάποια στοιχεία, να σας συνοψίσω και να σας δώσω την εικόνα του γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι ήταν το 2016 σημαντικό και θετικό έτος και από πλευρά ανάκαμψη τη οικονομία αλλά και καλών ρυθμών ανάπτυξη. Οι προσδοκίε στην αρχή του 2016 ε, έλεγαν ότι θα πάμε σε ανάπτυξη του 2%. Τελικά όμω φτάσαμε το 3% ρυθμό ανάπτυξη. Τα τελευταία πέσμα στοιχεία ε, λένε ότι το 2016 ε, φτάσαμε στην ε, κατά 2,9% αύξηση του ΑΕΠ. Βασικό στοιχείο σε αυτό ήταν η αύξηση των εξαγωγών. Οπότε και αυτό βοήθησε όσον αφορά το να σταθεί στα πόδια τη οικονομία μας. Ε, Βεβαίω βοήθησε και το ότι είμαστε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση πέραν των εξαγωγών. Ε, επίσης διαπιστώθηκε ότι έχουν αυξηθεί και οι εισαγωγέ. Επομένω υπήρξε εξουδετέρωση των εισαγωγών από τις εξαγωγές και αντίστροφα αύξηση τη κατανάλωση αλλά και των επενδύσεων. Οπότε κατόπιν σημαντικού χρονικού διαστήματος είχαμε επιτέλους όχι μόνο ανάκαμψη αλλά και σημαντικές επενδύσεις. Όσον αφορά τώρα την παραγωγικότητα, από όλους τους τομείς και κλάδους της οικονομίας είδαμε πολύ καλές επιδόσεις το 2016. Ξεκινούμε από την βιομηχανία. Ε, ανεβήκαμε από το 5% και όσον αφορά ε, <clears throat> τώρα τον τουρισμό που γνωρίζετε ότι είναι σημαντική δραστηριότητα για μας και 18 με 20% ήταν η συμβολή στο ΑΕΠ ετησίως. Επίσης θα πρέπει να σταθούμε σε μια άλλη δραστηριότητα που μετά από μια πτώση την τελευταία εξαετία ε, τώρα φτάσαμε σε θετικές ε, επιδόσεις. Μιλούμε για τις κατασκευές και όλες αυτές οι δραστηριότητες επομένως που προαναφέραμε τα πήγαν καλά ταυτοχρόνως θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τα Όπως και εσείς είπατε, ακριβώς διότι τα δημισιονομικά χειροτέρευσαν, ε, ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την διαδικασία που ονομάζεται EDP, για την ξεκίνησε για την Κροατία και το αποτέλεσμα ήταν στο να εξεταστούν διάφορες πλευρές της ε, δημοσιονομικής μας πολιτικής. Αναγνωρίσαμε για το ότι η χρηματοοικονομική μας θέση είναι βασική πρόκληση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αμέσως το πρόβλημα αυτό. Και βέβαια έχουμε καταφέρει τον τελευταίο 1,5 χρόνο που δεν είναι και ε, ε, πολύ καταφέραμε σε αυτό το σύντομο διάστημα να αντιστρέψουμε τις αρνητικές τάσεις και να πετύχουμε σημαντικά. Στην αρχή είχαμε κάποια ελλείμματα που ήταν 2,6% του ΑΕΠ. Ευθεία στήκαμε μετά με τις συστάσεις για την χώρα και επομένως ε, προσπαθήσαμε να εντάξουμε το έλλειμμά μας στα κριτήρια του Μάστριξ, δηλαδή να είναι κάτω από το 3%. Βέβαια είπαμε την τελευταία εξαετία τα ελλείμματα ήταν πάνω από 5% του ΑΕΠ. Παρ' όλα αυτά, για όλη τη χρονιά μπορέσαμε να ελέγξουμε τις δαπάνες και αξιοποιήσαμε τα πλεονάσματα των εσόδων για το έλλειμμα και τη συρρήκνωση του χρέους. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν τότε, τον Δεκέμβριο είχαμε συμπληρωματικό τεχνικό προϋπολογισμό λόγω της καινούργιας κυβέρνησης. Και από το 2,6 πήγαμε στο 1% του ΑΕΠ όσον αφορά τον στόχο για το έλλειμμα τον επόμενο δε μήνα. Πρόκειται να υποβάλουμε τους σχετικούς πίνακες στην Eurostat. Οπότε τότε θα δούμε όλοι τα νέα επίσημα στοιχεία. Αλλά μία πρόγευση είναι το εξή. Αυτό που σας είπα το 2016, αλλά για το συμπέρασμα ότι δεν είναι μόνο το θέμα του 1,6% του ΕΠ το οποίο καταφέραμε, αλλά το ότι πάμε ακόμα καλύτερα τώρα και ε, τελικά πάμε σε έλλειμμα 1% του ΑΕΠ. Επομένως, ανάπτυξη, εξυγίανση δημιουργικών και κατά τρίτον έχουμε την ε, δραστηριοποίηση της ε, περιουσίας του κράτους, των επιχειρήσεων δηλαδή, αλλά και άλλα πορτφόλιο για άλλα στοιχεία της ε, κρατικής περιουσίας ε, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ε, τουριστικές εγκαταστάσεις, όλα αυτά αξιοποιήθηκαν και έτσι όλα αυτά βοήθησαν στο ότι η χώρα μας για πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία της κατάφερε να συρρυκνώσει το ποσοστό του χρέους, 86,7% στο 84%, 83,9% τώρα και μάλλον θα, θα υπάρξει πτωτική τάση. Επομένως, ε, τελικά μειώθηκε από, το, από την κρατική προσπάθεια 3% το χρέος. Ε, επομένως, σε όλη αυτή τη δεκαετία τώρα καταλήξαμε σε αυτή την θετική κατάληξη. Βέβαια, ακόμα είμαστε δύο θέσεις ε, πιο κάτω από εκεί που πρέπει από πλευρά ε, των οίκων αξιολόγησης Fitch αλλά τέλος πάντων ε, εμείς θα συνεχίσουμε αυτή μας την πορεία και θα προχωρήσουμε τις διορθωτικές μεταρρυθμίσεις που είναι ότι έχει συσταθεί στη χώρα, ότι έχει ζητήσει η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, αλλά θα προχωρήσουμε και σε δράσεις και μέτρα που πιστεύουμε ακράδαντα ότι χρειάζονται και θέλουμε επομένως να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την μακρόπνοη βιωσιμότητα των οικονομικών μας επιδόσεων και, και δημιουργικών δημιουσιονομικών. Οπότε τώρα έχουμε κάποιους ε, στόχους μεσοπρόθεσμους. Αυτοί βεβαίως έχουν σχέση με τις δυνατότητες ανάπτυξης της οικονομίας. Καταφέραμε ακόμη περισσότερο όμως από αυτά, άρα και χρειάζεται να προσπαθήσουμε και να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τους ρυθμούς ε, των μεταρρυθμίσεων. Σύντομα πρόκειται να έχουμε το εθνικό πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων και, και σύγκλησης οπότε θα δείτε ποια είναι τα στοιχεία που αποτελούν ε, αυτές μας τις πολιτικές. Θα δείτε ότι προσπαθούμε για την υγεία, για τη διοίκηση, για τις συντάξεις, αλλά επίσης και στο μέτωπο του να βελτιώνουμε το επιχειρηματικό κλίμα και τις σχετικές δραστηριότητες. Θέλουμε και μπορούμε να τηρήσουμε αυτές μας τις υποχρεώσεις, τις υποσχέσεις, τις δεσμεύσεις για τις μεταρρυθμίσεις. Ήδη το απέδειξε αυτό η κυβέρνησή μας ευθύς εξ αρχής της εντολής μας. Υποβάλαμε προς ψήφι στο Κοινοβούλιο αυτή μας την ε, πολιτική και ξεκινήσαμε αυτή την ε, διαδρομή που αφορά την μεταρρύθμιση της ε, φορολογίας. Μιλούμε για 15 νομοθετήματα και 30 και πάνω δευτερεύοντα νομοθετήματα ε, για να προσπαθήσουμε να έχουμε απλούστευση του φορολογικού δικαίου, να είναι πιο αποτελεσματικό το φορολογικό μας σύστημα, να οδηγεί σε περισσότερη σταθερότητα την οικονομία της χώρας. Επίσης θα λάβουμε υπόψη ε, και κάποια άλλα στοιχεία ε, που θα αποτελούν φοροαπαλλαγές για ε, οικοκυριά και επιχειρηματίες μιλούμε για 7% του ΑΕΠ και αυτό θα αφορά κάποιους τομείς που θα διαπιστώσουμε ότι αφορούν αυτά τα σημεία ε, την οικονομική μας ανάπτυξη, δηλαδή τους φόρους ε, των εταιριών αλλά και εισοδήματος φυσικών προσώπων. Για τη δημοσιομική και γενικότερα για την οικονομία η βασική προτεραιότητα είναι το πώς θα απορροφούμε και θα αξιοποιούμε τους κινητικούς πόρους. Ακόμα και για τον προϋπολογισμό του 2016 νομίζω τα πήγαμε καλά. Αλλά μπορούμε να τα πάμε ακόμα καλύτερα και με τη βοήθεια των κοινωνικών κονδυλίων μπορούμε να δώσουμε συνέχεια ε, στις προσπάθειες για τις ε, υποδομές. Αλλά επίσης νομίζω ότι έτσι μπορεί να καταφέρουμε καλύτερα όσον αφορά την πραγματική οικονομία ή την οικοδομική δραστηριότητα. Τέλος πάντων, ευχαριστώ να απαντήσω σε σχόλια, σε ερωτήσεις. Αλλά όπως ε, σας είπα, τα πήγαμε πιστεύω καλά τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Έτσι δείξαμε, αποδείξαμε, μπορούμε να αντιστρέψουμε γρήγορα τις αρνητικές τάσεις. Όμως, έχουμε μπροστά μας μια σημαντική περίοδο πρέπει να συνεχίζουμε, πρέπει να επιταχύνουμε, να εντύρουμε τις προσπαθίες μας για τις μεταρρυθμίσεις. Και εκεί να καταφέρουμε τη χρήση για την ανάπτυξη, να έχουμε μια ισχυρή δημοσιονομική θέση, να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και στο μέτωπο της ε, σύγκλησης και σε με τους μέσους όρους που επιτάσσει η Σας, Σας ευχαριστώ για τις ε, πραγματικά πλήρες παρατηρήσεις σας. Νομίζω ότι Αυτά τα οποία είπατε θα έλεγα είναι πράγματα που χαρακτηρίζουν και αυτά τα οποία πολλοί που μας κατηγορούν να αναφέρουν το θέμα των διαφορετικών ανισορροπιών σαν παράδειγμα και πώς οι δείκτες ονομαστικού ελλείμματος μπορεί να βελτιώσουν ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου θέματα ελλείμματος και όταν μπείτε γρήγορα εύχομαι στο προληπτικό αν θέλετε κομμάτι τότε θα έχετε κάποιους στόχους που θα καθορίζονται από την γνωστή μετρική η μετρολογία καλύτερα των διαρθρωτικών μέτρων. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, αλλά, ελπίζω, αλλά είμαι σίγουρος ότι η περίπτωσή σας παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η κυρία Μάλετιτς είναι η πρώτη ομιλήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ Δράβκο, καλώ ήρθες στην ΕΚΟΝ. Χαίρομαι που είσαι μαζί μας σήμερα. Είσαι ο πρώτο υπουργό από την Κροατία που έρχεσαι ε, στα πλαίσια του διαλόγου με την Επιτροπή μας και γι' αυτό θα συνεχίσω την ερώτησή μου στην κροατική. Uvodno si jako dobro objasnio situaciju i čestitam na svim aktivnostima koje su poduzete vezano uz smanjenje duga i deficita, to je istaknuo i predsjednik našeg odbora. Zaista se vidi da se javnim financijama jako dobro i kvalitetno upravlja i da se ciljevi ispunjavaju.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 U isto vrijeme naravno da i iz perspektive proračuna, ali poglavito iz perspektive ukupne ekonomije i makroekonomije sigurno da su jako važne neravnoteže koje su identificirane od strane europskih institucija, ali tako isto od strane hrvatskih vlasti odnosno Vlade.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 Ευχαριστώ πολύ. Ο Σφεν Γίγολτ. thank you um, for, your Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα. Και θα ήθελα να θίξω το θέμα των συστάσεων αναχώρα. Στην περίπτωση πολλών χωρών, χωρίς να εξαιρείτε και η δική σας, ε, είδαμε οι συστάσεις αυτές να έχουν συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Είδαμε δηλαδή ότι κατά την αξιολόγηση του εξαμήνου η Κροατία το 2016 αντέδρασε με καθόλου ή με περιορισμένη πρόοδο το 2014, το 2015 σε πέντε συστάσεις δεν είχαμε καθόλου πρόοδο και σε μία σύσταση πολύ περιορισμένη πρόοδο. Σκοπεύετε να πάρετε πιο σοβαρά τις συστάσεις αυτές ή θεωρείτε ότι δεν είναι σκόπιμες. Η κυβέρνησή σας υπερψήφισε τις συστάσεις αυτές στο Συμβούλιο. Εγκρίνατε λοιπόν τις συστάσεις, αλλά υπάρχει περιορισμένη πρόοδος κατά την εφαρμογή τους. Και μήπως μπορείτε να μας ε, εξηγήσετε ένα θέμα που μου φαίνεται κρίσιμο σε πολλά κράτη-μέλη. Το θέμα ότι το δικαστικό σύστημα δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό και θα πρέπει να λαμβάνει πιο γρήγορα αποφάσεις. Μήπως ε, μπορείτε να μας αναπτύξετε περισσότερο τα σχέδια σας σχετικά με τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, όπως αναφέρετε στις συστάσεις αναχώρα. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και παρατηρήσεις σας. Οπωσδήποτε θα απαντήσω στην ερώτησή σας. Παίρνουμε απολύτως στα σοβαρά τις συστάσεις αναχώρα και όχι μόνο επειδή προέρχονται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και λόγω του ότι συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με τους δικούς μας προβληματισμούς ως κυβέρνηση. Ο λόγος που είχαμε περιορισμένη ή καθόλου πρόοδο, ιδιαίτερα το 2016, Αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο είχαμε δύο κοινοβουλευτικέ εκλογέ. Ε, Τι κανονικέ στο τέλος του 2015, που είχαν ως αποτέλεσμα τρεις ε, ή τέσσερις μήνες σχηματισμού της κυβέρνησης. Μετά από έξι μήνες από το σχηματισμό της κυβέρνησης έπεσε πάλι η κυβέρνηση και είχαμε πάλι εκλογές. Αυτό λοιπόν ήταν σημαντικός παράγοντας καθυστέρησης ε, στις συστάσεις αναχώρα. Όπως όμως ε, θα γνωρίζετε, καταφέραμε να κρατήσουμε υποέλεγχο τα δημοσιονομικά και έτσι περιμένουμε τον ε, Μάιο έξοδο από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Επίσης, ε, τον ε, Μάιο θα ε, επισημάνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του μίσο που βλέπουμε να έχει σημειωθεί πρόοδο όσον αφορά τι ε, διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει. Ε, και οι μεταρρυθμίσει αυτέ ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με τι συστάσει αναχώρα. Και είτε μιλάμε για το επιχειρηματικό περιβάλλον, το σύστημα υγεία ή και το θέμα που θίξατε εσεί, το δικαστικό δίστημα δηλαδή και το νομικό μα πλαίσιο Είμαστε αρκετά σαφείς. Και όπως απάντησα και στην προηγούμενη ερώτηση του Ιβαν Μάλετης, θέλουμε να βελτιώσουμε το δικαστικό μας σύστημα, όχι μόνο για να υπάρχει περισσότερη σταθερότητα, αλλά να υπάρχει και συνέπεια και προβλεψιμότητα και επίσης να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος όσον αφορά τον σεβασμό του κράτους δικαίου και την προστασία και όσων επενδύουν στη χώρα μας. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα στοιχείο κλειδί, ώστε η Κροατία να γίνει πιο ελκυστικός τόπος για επενδύσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπάνεμαντς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εάν κατάλαβα σωστά, κύριε Υπουργέ, Θέλετε πολύ να προσχωρήσετε στην Ευρωζώνη. Υπάρχουν όμως πολλές δυσκολίες στην Ευρωζώνη. Η κυβέρνησή σας δεν ανησυχεί σχετικά με τη σταθερότητα στην Ευρωζώνη. Τι γίνεται με τους πολίτες. Είναι δύσκολο να σας κάνω παρατηρήσεις, αλλά διάβασα στο Ευρωπαρόμετρο ότι το μισό των Κροατών πολιτών ε, βλέπουν αρνητικά την προσχώρηση στο ευρώ. Η κυβέρνησή σας, ε, λοιπόν, πώς το βλέπει αυτό. Διστάζει καθόλου με βάση τις πληροφορίες αυτές του Ευρωβαρόμετρου. ή προβλέπετε να, είσαστε, να συμμετέχετε με άλλο τρόπο όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, σας ευχαριστώ πολύ και για την ερώτηση και για την παρατήρησή σας. δύο γεγονότα να σας αναφέρω. Πρώτο απαντήσω, διότι ιστορικά η Κροατία είναι πολύ ευρωπαϊκή οικονομία, συνδέεται στενά με την γερμανική οικονομία πάνω από το 70% και στις δύο πλευρές του ισοζυγίου συνδέονται με την Ευρώπη. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Το άλλο, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι το γεγονός ότι με την προσχώρησή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αναλάβαμε ως υποχρέωση να εισάγουμε το ευρώ. Για να γίνει αυτό όμως ε, πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Και απαιτούνται και πολιτικές αποφάσεις. Η Κροατία αυτή τη στιγμή πληρεί 4 στα 5 κριτήρια. Το μόνο που δεν πληρούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι παρότι μειώθηκε το 2016 για πρώτη φορά ε, το, ε, το δημόσιο χρέος, ε, παραμένει στο 60%. Όπως είπα και πριν όμως, στο έγγραφο που υιοθέτησε πριν δύο μήνες η κυβέρνηση σχετικά με τη στρατηγική για το δημόσιο χρέος, Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε ε, την μείωση του δημοσίου χρέους ε, κατά 2,5 με 3% κάθε χρόνο, κάτι που ευθυγραμμίζεται με το Σύμφωνο Σταθερότητας, καθώς ε, και με όλους τους άλλους κανονισμούς που λένε ότι ακόμα και αν έχει ξεπεράσει κανείς το 50% θα πρέπει να αναθεωρεί προς τα κάτω το δημόσιο χρέος κατά 20% και Η Κροατία αυτή τη στιγμή πληρώνει περίπου το 3,5% ε, του ΑΕΠ σε τόκους. Αυτό σημαίνει ότι είχαμε πρωτογενές πλεόνασμα άνω του 2% του ΑΕΠ. Όσον αφορά την εισαγωγή του ευρώ, παίρνουμε πολύ στα σοβαρά την παρατήρησή σας και όχι μόνο τη δική σας παρατήρηση, αλλά φυσικά και τη γνώμη των πολιτών μας σκοπεύουμε μαζί με την Εθνική μας Τράπεζα να κάνουμε μια εντελεχή ανάλυση κόστους-όφελους, κάτι που δεν έχει γίνει εδώ και κάποια χρόνια στην Κροατία. Σίγουρα παρακολουθούμε τις τάσεις στην Ευρωζώνη, καθώς και τις εξελίξεις σε σχέση με το Brexit. Στην ανάλυση κόστους-όφελους θέλουμε να έχουμε ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων που συνδέονται με την εισαγωγή ή όχι του ευρώ. Αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να λάβουμε τελικά την αποφασή μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι βέβαιος Ε, ότι θα λάβετε υπόψη σας και τα δάνεια σε ελβετικά φράγκα κατά την ε, ε, απόφασή σας αυτή. Ευχαριστώ κύριο Μάιερ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που βρίσκεστε εδώ πέρα και απαντάτε ευγενικά στις ερωτήσεις μας. Έχω τρεις σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με την οικονομική ανάπτυξη. Στα δεδομένα βλέπω ότι η χώρα σας ανακύπτει από το 2012 έως το 2015 βρισκόσασταν πίσω σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΑΕΠ κατά κεφαλήν είναι κάτω από το μέσο όρο, ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι γι' αυτό και πώς βλέπετε όλη την κατάσταση στην περιφέρειά σας, ε, κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Κοινοβουλίο μας. Όσον αφορά το δημοσιονομικό σχέδιο, θα πρέπει να σας συγχαρώ για την πρόοδο που έχετε σημειώσει. Δεν είναι εύκολο υπό τις προϋποθέσεις αυτές να ελέγξει κανείς τον προϋπολογισμό, ε, από την άλλη βλέπω ότι στα επόμενα χρόνια ε, σκοπεύεται να ε, διευρύνεται το έλλειμμα και επίσης και εγώ και κάποιοι συνάδελφοι που δεν είναι παρόντες εδώ θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι ισχύει όσον αφορά τον νόμο για τη μετατροπή σε ευρώ και φράγκα κάτι που θεωρήθηκε οριακό όσον αφορά την νομιμότητα. Ε, ευχαριστώ. Όσον αφορά την ερώτησή σας ε, για το ΑΕΠ, μετά το 2,9 το 2016, ε, προβλέπετε το 3,2% για το 2017 και είμαι περήφανος που μπορώ να σας πω ότι και οι δικές μας προβλέψεις είναι σχεδόν όμοιες με της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλων των σχετικών οικονομικών Ινστιτούτων και ε, οικονομολόγων. Ε, είτε μιλάμε για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είτε μιλάμε για εγχώριους. Ε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει 3,1% ανάπτυξη. Όπως είπα και στην εισαγωγή μου, μετά από μακρά περίοδο ύφεση και μείωση του ΑΕΠ, με συνέπεια μείωση το κατακεφαλήν ΑΕΠ, η ανάπτυξη και η μείωση του ελλείμματος ε, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για μας. Ε, θέλουμε να μπούμε στο δρόμο της σύγκλησης ε, και να φτάσουμε την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο όσον αφορά τον μεσόρο, αλλά και όσον αφορά τις τάσεις. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελευταία πρόβλεψή της θεώρησε την Κροατία μία από δύο χώρες όπου είχαμε αναθεώρηση προς τα πάνω. Αυτό Σαφώς είναι σαφής απόδειξη ότι έχουμε μεγάλο βαθμό αναγνώρισης των ε, μέσων και των δράσεων που σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε. Όσον αφορά τη δημοσιονομική μας θέση, νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας όσον αφορά ε, το διαρθρωτικό έλλειμμα. Ωστόσο, πρέπει να το απαντήσω αυτό λέγοντας ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και το 2016 και το 2017 το 2016 αποδείχθηκε πολύ πολύ καλύτερο από ό,τι αναμενόταν αρχικά. Και ε, η πρόοδος ε, όχι μόνο ξεπερνούσε τις ε, προσδοκίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, αλλά και τις δικές μας προσδοκίες κατά την εκπόνηση του προπολογισμού για το 2017. Ε, ο στόχος ε, ήταν να έχουμε ανάπτυξη 1,6 έως 2% και το 2017 να έχουμε περαιτέρω προσαρμογές. Τώρα με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε για το 2016 έχει αποδειχθεί ότι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Ωστόσο για το 2017 μπορώ να σας πω ανοιχτά και ειλικρινώς ότι θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε την ίδια στρατηγική για τα δημοσιονομικά και το κλειδί της επιτυχίας μας βρίσκεται στην πλευρά των δαπανών. Σε αυτόν τον τομέα πρέπει να έχουμε καλό έλεγχο, πιο ορθολογιστική χρήση των ε, δημοσίων πόρων και στρατηγική για τη μείωση του χρέους. Αυτή λοιπόν ε, είναι η στρατηγική μας σήμερα. Ναι, βρισκόμαστε ακόμα στο πρώτο τρίμηνο του 2017. Ε, μας περιμένουν πολλές προκλήσεις το έτος αυτό, αλλά ο στόχος μας είναι να βελτιώσουμε το, τον ισολογισμό μας και όσον αφορά το ελβετικό φράγκο, ε, έχουμε ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πριν το καλοκαίρι, το συνταγματικό μας δικαστήριο θα λάβει απόφαση στην ε, εν λόγω υπόθεση και θα συνεχίσουμε το διάλογό μας. Ε, καταλαβαίνουμε πολύ καλά το πλαίσιο και ε, τα βασικά επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την υιοθέτηση του νόμου αυτού. Πάνω από το 94% των οφηλετών που είχαν στεγαστικά δάνεια σε ελβετικά φράγκα τα μετέτρεψαν το οποίο σημαίνει ότι είναι πολύ μικρή η πιθανότητα να χρειαστεί να εφαρμοστεί, ωστόσο έχουμε προορατική προσέγγιση και διάλογο με τις τράπεζες στην Κροατία και συζητάμε διάφορες δυνατότητες και επιλογές για να μπορέσουμε να βρούμε μια ικανοποιητική λύση αμοιβαία αποδεχτή που να μην διακυβεύει τη δημοσιονομική μας θέση. Και κάτι το οποίο θα αποτελέσει αμοιβαία αποδεχτή λύση χωρίς να χρειαστεί να προσφύγουμε σε διατησία. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρος βέβαια, και πρέπει να ετοιμαστούμε για την επόμενη ερώτηση, αλλά θα είτε πάτε πολύ. Γι' αυτό και κόμπρον, για το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Μάριτς. Βεβαίω και η χώρα σα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρω. Αλλά όχι στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, στην Ευρωζώνη και η νομισματική σα πολιτική. Πάντοτε αυτή ενισόταν με το ευρώ. Αλλά θέλετε από το 2019 και μετά μέχρι το ευρώ. Όμως τι γίνεται με την ανεργία. Είναι 11,3% τον Ιανουάριο φέτος. Ακριβώς όπως Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία. Και οι νέοι έχουν ανεργία στο 40%. Όπως η Ισπανία, η Ελλάδα. Άρα ευθυγραμμίζεται σε αυτό το μέτωπο με τις νότιες ευρωπαϊκές χώρες. Αλήθεια, θέλετε να μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά όλη αυτή την ανεργία. Και θα δεχθείτε πρόγραμμα λιτότητας όπως αυτό που επευλήθη στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι η χώρα σας μπορεί να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστική μέσα στην ΟΝΕ και κυρίως θα δεχθεί ο λαός την λιτότητα. Και κοιτάξτε, τι γίνεται στην Ελλάδα. Καταστροφή, ταραχές στους δρόμους και όλα τα άλλα. Μα γίνονται αυτά στη χώρα σας, θέλετε να γίνουν. Είναι προς το συμφέρον σας. Εδώ δεν θέλουν να βγουν από το ευρώ. Α, η Ιταλία, ας πούμε. Thank you for your, uh, question. Ευχαριστώ και την ερώτησή λέει ο κύριος Να σας πω, εν συντομία, όπως και για την προηγούμενη ερώτηση που ετώνησα, ότι οπωσδήποτε θα κάνουμε προσεκτική ανάλυση κόστους ωφέλους και από όλες τις οπτικές γωνίες. Όλα τα υπέρ και τα κατά θα τα σταθμίσουμε για να μπούμε στην Ευρωζώνη. Και θα δούμε τι θα ισχύσει και για τα κέντρα αποφάσεων στη χώρα αλλά και για τον κόσμο. Τι ωφέλη υπάρχουν, τι απειλές, τι προβλήματα εάν υιοθετήσουμε το ευρώ. Αυτή είναι η επίσημη θέση προς το παρόν και στο άμεσο μέλλον βέβαια θα παρακολουθούμε τις ε, εξελίξεις τι θα γίνει στο Brexit τι θα γίνει στην Ελλάδα και όλα αυτά θα είναι μεταβλητές για να αποφασίσουμε Τώρα για την ανεργία που σχολιάσατε ιδίως όσον αφορά τους νέους για μας αυτό είναι μακράν το πιο σημαντικό στοιχείο για την οικονομική μας πολιτική και για την κυβέρνησή μας πιο σημαντικό στοιχείο από το, ρυθμό της ανεργίας, ποσό της ανεργίας είναι το ποσό της απασχόλησης. Γι' αυτό και πάμε για μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας. Σε αυτό το μέτωπο θέλουμε να ρίξουμε το βάρος μας και τις προσπάθειές μας και σε σχέση και με την ισοτιμία όπως είπατε είναι και το θέμα της συνταγωνιστικότητας και από τότε που το 1934 υιοθετήσαμε το Κούνα η κοινική Τράπεζα ε, ακολουθεί μια πολύ σφιχτή πολιτική ισοτιμιών με πάρα πολύ μικρό περιθώριο διακύμανσης. Οπότε έχουμε πετύχει την τελευταία 25 ετία μια καλή επίδοση. Βεβαίω και έχουμε τον προβληματισμό του ε, πώ μπορούμε να κερδίσουμε σε ανταγωνιστικότητα με κάποιο είδο ονομαστική υποτίμηση κλπ. Αλλά τέλο πάντων το συμπέρασμα το κλασικό είναι ότι θα πρέπει να γίνει εσωτερική υποτίμηση του νομίσματος. Αν είναι να γίνει. πλέον να αναφέρατε και τη λιτότητα και τα λοιπά που συνδέονται με αυτήν. Το 2016 μπορώ να σας πω ότι φάνηκε ξεκάθαρα πώς κανείς μπορεί να είναι υπεύθυνος διαχείρισης των νομικών Γιατί είχαμε πάγωμα της δημόσιας δαπάνης για πρώτη φορά και χρησιμοποιήσαμε το πλεόνασμα και τα έσοδα και γι' αυτό και μειώσαμε και τις τρύπες στο ΕΠ. Και νομίζουμε ότι αυτή είναι η καλύτερη συνταγή εξυγίανσης και σταθερότητας των δημοσιονομικών. Έτσι πρέπει κανείς να βαδίζει. Α, εκεί κατευθύνουμε τις προσπαθίες μας. Ο κύριος ο επόμενος από τη Ρουμανία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Ιβάν να σας μιλήσω στην μητρική μου γλώσσα και πρώτα πρώτα συγχαρητήρια για την πρόοδο που πετύχατε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι πολύ καλά τα μαντάτα από πλευρά τη οικονομική πολιτική. Οπότε και είναι ρητορικό το ερώτημα τελικά. Το εάν θα τα πηγαίνατε το ίδιο καλά, εάν βρισκόσασταν στην Ευρωζώνη. Διότι πολλά από τα εργαλεία που μετήλθατε κατά αυτή την περίοδο δεν θα τα είχατε εάν ανήκατε στην Ευρωζώνη. Ε, τελικά το να μπήκαν στην Ευρωζώνη όχι είναι θέμα τεχνικό, οικονομικό, δεν είναι πολιτικό. Ε, αυτά τα έχουμε πει και για άλλες χώρες που είναι να μπουν στην Ευρωζώνη. Αλλά για πετε μας. Θεωρείται από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σωστό το ότι κινούνται μόνο προς το να σέψουν τον πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα έπρεπε να κάνουν κάτι και για την ε, απασχόληση όπως ακριβώς κάνει και η Κεντρική Τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν τα κάνει αυτά η Καπατάφ. Μάριτ, σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Για να είμαι ειλικρινής, πρώτη φορά κάποιος μου ζητάει να σχολιάσω τα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μα θέμα είναι τι κάνει δική μας Κεντρική Τράπεζα. Πάντως, Αυτά τα οποία λέω προς τη δική μας κεντρική τράπεζα θα τα έλεγα και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή ως Υπουργό Οικονομικών αλλά και ως Οικονομολόγο, πιστεύω ότι ο στόχος δεν είναι μόνο η σταθεροποίηση των τιμών. Αυτό βέβαια είναι θέμα νομισματικής πολιτικής αλλά και φορολογική πολιτική. Θα πρέπει κανεί να προσέχει την οικονομική δραστηριότητα, θα πρέπει κανεί να δουλεύει και για την ε, απασχόληση, όπω είπαμε και στο προηγούμενο ερώτημα. Θα πρέπει κανεί να βρίσκει το κατάλληλο policy mix μεταξύ των ε, επιμέρους οικονομικών μετόπων και να βρει με ποιε συνταγέ θα, θα αναβαθμίσει την οικονομική δραστηριότητα, θα βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο, αλλά και θα βελτιώσει την κατάσταση στην αγορά εργασίας. Ε, πολύ σημαντικό αυτό και στη δική μας περίπτωση έχουμε καλή σχέση με την κεντρική τράπεζα της χώρας. Και βέβαια είναι βασικά μες οι αρμοδιότητες μας για το τι μπορούμε να κάνουμε από πλευράς αυτής. Πάντως, χρειάζεται κανείς να έχει μια πολιτική που στοχεύει και προς τα συγκεκριμένα προβλήματα αλλά και γενικότερα προς την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης. Η κυρία Μάλετιτς. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω ε, κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει προγνωστικά, αναλύει, συστήνει και απευθύνει σε διάφορες χώρες. Χρειάζεται βέβαια όμως να υπάρξει πρόσβαση σε δανεισμό από πλευράς των επιχειρηματιών. Να υπάρχει επίσης βοήθεια προς την έρευνα και ανάπτυξη. Όμως για την Κροατία δεν προσφέρονται τόσο πολλές τέτοιες δυνατότητες. Μικρές οι επενδύσεις, μικρά τα χρηματικά ποσά. Άρα ακόμα δεν βοηθάται όσο πρέπει η πραγματική οικονομία. Γι' αυτό και έχουμε τόσο πολλά κόκκινα δάνεια. Για πέστε μας, τι στρατηγική έχετε ως προς αυτό. Να σας τα πω στα αγγλικά, λέει ο κύριος Μάριτς, όπως μας είπατε. Το επίπεδο των NPL, των κόκκινων δηλαδή των μη εξυπηρετούμενων δανείων, στο τέλος του 2016 άρχισαν να μειώνονται τα ποσοστά τα οποία είχαμε, είναι γύρω στο 50% αν συγκρίνουμε με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στον τομέα του επιχειρηματικού δανείου, ε, θα πρέπει να πάρουμε δράσεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Εμείς το αναγνωρίζουμε αυτό και στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων των φορολογικών και στα πλαίσια του καθορισμού του πεδίου επιβολής ε, του ε, φόρου επί των επιχειρήσεων. Προσπαθούμε να δώσουμε κίνητρα στην ε, χρηματοπιστωτική ή γενικά πλευρά έτσι ώστε να δείξουν μεγαλύτερη, θα έλεγα, ικανότητα διαχείρισης των NPL όχι μόνο για να διευρυνθούν οι δυνατότητες έβρεσης πηγών ρευστότητα για τις επιχειρήσεις, αλλά και ε, να μπορέσουν να απελευθερωθούν λίγο από την απλή διαχείριση των κόκκινων δανείων ε, και να μπορέσουν να ασχοληθούν γενικά με την οικονομική ε, δραστηριότητα και ανάπτυξη. Φυσικά ο τραπεζικός τομέας highly liquid. We are having overnight deposits on market, which is in range between... Οι χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και οι πιστωτικές δραστηριότητες στη χώρα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, διασφαλίσουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ρευστότητας της χώρας και έχουν και ένα ποσοστό κάλυψης κεφαλαίων, αν ακούσαμε καλά, γύρω στο 20% όλα αυτά διστάζουν να διαθέσουν τα ε, κεφάλαια τα οποία έχουν στη διάθεσή τους γιατί ακριβώς υπάρχουν πάρα πολλά NPL ε, ε, στις αγορές και γι' αυτό θα πρέπει να αλλάξει η κατάσταση. Ελπίζω αυτό να γίνει με τα καινούργια μέτρα και επανέρχομαι εδώ και στα ευρωπαϊκά ταμεία τα οποία είναι καθοριστικός παράγων χρηματοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων όπως η υγεία, η επιστήμη, η εκπαίδευση και κανονικά θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ποσά αυτά από τους πόρους τους εσωτερικούς τους οποίους διαθέτει η χρηματοπιστωτική δραστηριότητα στη χώρα μου. Και μια τελική παρατήρηση είναι ότι μία από τις βασικές δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουμε σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες είναι το χαμηλό επίπεδο κεφαλαιοποίησης των επιχειρήσεών μας. Γι' αυτό λοιπόν πέρα από το τι χρειάζεται να γίνει σε επίπεδο τραπεζών θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και σε επίπεδο ιδίων κεφαλαίων ε, των ε, επιχειρήσεων της χώρας. Η ύφεση οικονομική στη χώρα μου κράτησε πάρα πολλά χρόνια και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει προβλήματα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γουλφ, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Υπουργέ. Ήταν ε, χρήσιμο που ακούσαμε και την αισιοδοξία σας για την οικονομική πορεία της χώρας. Είχα μια ερώτηση σχετικά με την ανεργία, την έθεσε ο κύριος Κόμπερν. Η επόμενη ερώτηση, πέρα από το ποσοστό αυτό ανεργίας 11,3% γενικό ποσοστό και 43% σε επίπεδο ανεργίας νέων, είπατε ότι πέρυσι πετύχατε οικονομική ανάπτυξη σημαντική. Υπήρξε αύξηση της δραστηριότητας στον τομέα της οικοδομής και των εσόδων από τουρισμό. Ίσως αυτό να είναι λίγο παραπλανητικό. Μήπως πρέπει να πούμε ότι η ανάπτυξη του ΑΕΠ ε, προήλθε και από άλλα δύο θέματα στα οποία δεν αναφερθήκατε. Το πρώτο και το λέει η Παγκόσμια Τράπεζα είναι ότι η αύξηση χρηματοδότησης από το ΔΝΤ την Παγκόσμια Τράπεζα ε, το ΔΝΤ έχει φτάσει σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα του ε, προϋπολογισμού σας. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και μια δεύτερη πλευρά που εξηγεί το γιατί πετύχατε τα ποσοστά στα οποία αναφερθήκατε είναι ότι ιδιωτικοποιείται ε, περιουσία εθνική πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν. Και νομίζω ότι οι δύο αυτοί παράγοντες δείχνουν ακριβώς το ίδιο σενάριο το οποίο επευλήθη στην Ελλάδα πριν εισέλθει στο ευρώ. Αναφερθήκατε και στο Brexit και πρέπει και εγώ να αναφερθώ σε αυτό. Εσείς βλέπετε την εξέλιξη της οικονομίας σας μακροπρόθεσμα. Βλέπετε ότι υπάρχουν εξαιρετικοί παράγοντες που επηρεάζουν τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ε, θα χτυπήσουν και τη δική σας χώρα και ένα από τα προβλήματα είναι το Brexit. Έχει προετοιμαστεί η κυβέρνησή σας για μία μελέτη επιπτώσεων σε σχέση με το ΑΕΠ, με τις εξαγωγές, με τον τουρισμό. Τι θα συμβεί με τη μείωση σαν παράδειγμα των διαρθρωτικών ταμείων και μια τέτοια αξιολόγηση την έχετε μεταφέρει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή και στο ίδιο το Eurogroup. Σας ευχαριστώ. Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω με όλα τα δεδομένα τα οποία μας είπατε και σε σχέση με το ΑΕΠ, πέρα από την εσωτερική ζήτηση η οποία ήταν ο καθοριστικός παράγων της συμπεριφοράς μας σε επίπεδο ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν φυσικά και άλλοι παράγοντες οι οποίοι είναι εξωγενείς. Οφεληθήκαμε επίσης και από τις χαμηλές τιμές των καυσίμων, και επίσης και κάποια προγράμματα διευκόλυνσης σε επίπεδο ρευστότητας έχουν βοηθήσει την οικονομική μας επίδοση τον προηγούμενο χρόνο. Αυτό όμως έχει σχέση και με την υψηλή ανθεκτικότητα της κορατικής οικονομίας. Ο τουρισμός, σαν παράδειγμα, συμμετέχει κατά 18 με 20% του ΑΕΠ της χώρας των εσόδων συγγνώμη, της χώρας. Ο τουρισμός λοιπόν έχει επιδείξει ότι είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός. Αυτό οφείλεται και στο ότι οι ανταγωνιστές μας σε μεσογειακές περιοχές αντιμετωπίζουν άλλου είδους προβλήματα. Πάντως, ιδιαίτερα στον ξενοδοχειακό τομέα, οι βασικοί πρωταγωνιστές εσωτερικοί και εξωτερικοί, παλαιοί και νέοι, είναι ισχυρότατη σε επίπεδο επενδύσεων. Και αυτό συνδέεται και με κάτι το οποίο είπατε σχετικά με την πώληση της δημοσίας περιουσίας. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει στην κατοχή της δεκάδες αλυσίδες ξενοδοχείων. Όχι γιατί θέλουμε εμείς να απαλλαγούμε από αυτά, αλλά στο παρελθόν λόγω πολλαπλών αλλαγών ιδιωτησίας κατέληγαν ε, στη φορολογική διοίκηση ε, σαν εγγύηση αν θέλετε και παρέμενε στην δημόσια σφαίρα. Και είναι αλυσίδες οι οποίες γενικά γίνονται αντικείμενο ε, τελούς θα έλεγα επιχειρηματικής διαχείρισης και γι' αυτό θα πρέπει να τα δραστηριοποιήσουμε ακόμα περισσότερο με τον ένα τρόπο ή τον άλλο, να βελτιώσουμε τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας γιατί από τη μία έχουμε στρατηγικούς επενδυτές, όχι απλούς χρηματοδότες, οι οποίοι ε, δίνουν την δυνατότητα μέσω των επενδύσεών τους να αυξηθεί το διαθέσιμο κεφάλαιο, να βελτιωθούν τα ξενοδοχεία, να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας και επίσης ε, να επηρεάσουν θετικά το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας τοπικά γύρω από τις μονάδες αυτές. Γι' αυτό λοιπόν επιμένουμε εμείς ε, στην ε, ε, δυνατότητα εκμετάλλευσης αυτής της περιουσίας για την ενίσχυση της, ευρωπαϊκής, της οικονομικής ολοκλήρωσης. Για το Brexit φυσικά και παρακολουθούμε από πάρα πολύ κοντά τις εξελίξεις, όχι μόνο σε επίπεδο Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά προσπαθούμε να αναλύσουμε και όλες τις άμεσες και κυρίως έμεσες συνέπειες. Όταν μιλάμε για το Brexit, ας πούμε, σε σχέση με τις εισαγωγές-εξαγωγές, γνωρίζετε ότι η Κροατία είναι πάρα πολύ χαμηλά σε σχέση με τις εμπορικές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα τελευταία δύο χρόνια, ένα-δύο χρόνια έχουν υπάρξει ε, αρκετές αυξήσεις, σαν παράδειγμα στον τουρισμό από τη χώρα σας. Και αυτό δεν είναι κακό αλλά νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν θα μας δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα και δεν θα θεωρηθεί σαν σημαντικό θέμα. Έμεσα όμως μπορεί να υπάρχουν προβλήματα και σε επίπεδο κεφάλαια αγορών θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τις συνέπειες και συνειδητοποιούμε πλήρως ότι οι συνέπειες αυτές. Η Περβάνς έχει το λόγο ξανά. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Αναφερθήκατε και εσείς στο Brexit. Οι ηγέτες μας μόλις οι πολιτικοί επέστρεψαν από τη Ρώμη και αναφέρθηκαν στο μέλλον της Ευρώπης των 27 χωρών. Ο συνάδελφος από τη Ρουμανία σας έθεσε ερωτήσεις για την ένταξή σας στη ζώνη ευρώ. Είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργεί προβλήματα στους 27 μήπως θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα θέματα που αφορούν το σύνολο των 27 ή να ασχοληθούμε ειδικά με το ευρώ. Στη δήλωση της Ρώμης υπάρχουν δύο αναφορές, άλλοι κρίνουν καλές, άλλοι άσχημες, σχετικά με την ενίσχυση του ενιαίου νομίσματος και ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Εσείς λοιπόν σαν μέλος του ΕΚΟΦΗΝ πώς βλέπετε να ολοκληρώνονται αυτές οι μελλοντικέ κινήσεις και κάτω από ποιες συνθήκες και κάτω από ποιο ρυθμό θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε παράλληλα και με τον Brexit και με την ολοκλήρωση της ε, ε, ε, νομισματικής αγοράς. Ανεξάρτητα αν είμαστε στην Ευρωζώνη ή όχι. Έχετε δίκιο. Προφανώς ε, στις συνεδριάσεις ΕΚΟΦΗΝ συζητάμε στοιχεία που συνδέονται όχι μόνο με το Brexit αλλά και με την ολοκλήρωση της νομισματικής ένωσης. Ο τρίτος πυλώνας είναι η εισαγωγή των, ε, του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων και Κατά τις συνεδριάσεις μας έχουμε πολύ αναλυτική συζήτηση, ιδιαίτερα με τις χώρες της Ευρωζώνης. Η Κροατία δεν συμμετέχει αυτή τη στιγμή σε αυτές τις ε, συζητήσεις, ε, αλλά λαμβάνει γνώση όλων των ε, πληροφοριών και παρακολουθεί τις εξελίξεις. Προφανώς, όλοι περιμένουμε την επίσημη έναρξη της διαδικασίας διαπραγματεύσεων, που αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα. Και μαζί με μια επαρκή βάση θα έχουμε καλύτερη σαφήνεια σχετικά με τα επόμενα βήματα. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει να απαντηθούν σύντομα για να μπορούμε να επιχειρηματολογούμε καλύτερα όσον αφορά το ερώτημα που θέσατε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Οικονομικών. Να σας συγχαρώ επίσης. Ήταν πολύ χρήσιμη επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Ευχόμαστε λοιπόν ό,τι καλύτερο στα επόμενα βήματα διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όσον αφορά την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και όσον αφορά την εφαρμογή των ε, αναχώρα συστάσεων. Επρόκειτο για την πρώτη μια ε, σειρά επικοδομητικών επαφών που θα έχουμε ανάμεσα στην Επιτροπή μας ε, και την κυβέρνησή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, παραδίδω την Προεδρία στον Μάρκους Φέρμπερ. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι η πρόταση οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με τους συντελεστέ του φόρου θέμενης αξίας για βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά. Είναι χαρά μου να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον Τόμ Φάντεν Καντελάρε. Here I am. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με την πρόταση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να βελτιώσει την παρούσα κατάσταση όπου τα κράτη-μέλη μπορούν να εφαρμόσουν μειωμένους ή πολύ μειωμένους συντηλιστές φόρου σε ε, βιβλία και τέτοια που δημοσιεύονται, όχι όμως ε, σε ό,τι δημοσιεύεται ηλεκτρονικά. Ε, η πολυ μειωμενους συντηλιστες φορου σε βιβλια και τετοια που δημοσιευονται οχι ομως σε οτι δημοσιευεται ηλεκτρονικα αρχικός στόχος ε, της, ε, της ε, πρότασης ήταν να διευκολυνθεί η κατάσταση, αλλά δεν αντικατοπτρίζει πια την πραγματικότητα σήμερα. Δεν πρέπει πια να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα έντυπα και τα ηλεκτρονικά δημοσιεύματα και ε, αυτό το πιστεύουν και τα πολλά κράτη-μέλη και εγώ. Υπάρχει το σχέδιο δράσης για το ΦΠΑ και γνωρίζουμε ότι το θέμα αυτό έχει οδηγήσει και σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις. Κατά τη γνώμη μου, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουμε μπροστά μα σήμερα είναι ισορροπημένη και δίνει την δυνατότητα στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν χαμηλού ή πολύ χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ στι ε, ηλεκτρονικά παρεχόμενε δημοσιεύσει. Ε, πρόταση αυτή νομίζω ότι έπρεπε ήδη να έχει εφαρμοστεί, θα πρέπει να υιοθετηθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και γι' αυτό επικροτώ την προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που διαχωρίζει την πρόταση αυτή από το γενικότερο καθεστώ ΦΠΑ. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη πρόταση έχει να κάνει με την ε, στρατηγική τη ενιαίας αγορά, λαμβάνοντα υπόψη την πραγματικότητα στι ψηφιακές οικονομίες που ζούμε σήμερα. Ακριβώ για τον λόγο αυτό ε, έχω ε, επιδιώξει ε, ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα, καθότι το Κοινοβούλιο επανειλημμένα έχει ζητήσει να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Ελπίζω γρήγορα να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε λύση. Αυτό αποτελεί και μήνυμα προς το Συμβούλιο, να επιταχύνει και εκείνο και να μην χρησιμοποιήσει το θέμα αυτό ως ε, διαπραγματευτικό εργαλείο για να πετύχει τη θέση του σε άλλα θέματα. Πιστεύω ότι το καθεστώς ΦΠΑ που περιμένουμε θα πρέπει να ε, αυξήσει την ευελιξία και να βελτιώσει το συντονισμό εντός μιας ε, ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Επίσης, ε, προσβλέπω σε ομαλή συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές. Σε ευχαριστώ, Τόμ. Δίνω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή, Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να προσθέσω σε αυτό. Η πρόταση αυτή είναι χρήσιμη, καλοδεχούμενη, δεν είναι πια λογικό να υπάρχει μείωση του ε, επίπεδου του συντελεστή του, στα έντυπα, να μην εφαρμόζεται επίσης και στις ηλεκτρονικές εκδόσεις. Η κατάσταση λοιπόν αυτή, θα έλεγα μέσω αυτής της πρότασης, ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει. Το θέμα δεν είναι η μορφή ε, ενός έργου, αλλά το περιεχόμενο του. Νομίζω ότι τα επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αρκετά για να μην υπάρξει επιβράδυνση της ε, διαδικασίας και διευρύνεται ουσιαστικά η ρύθμιση η οποία ισχύει στον συγκεκριμένο τομέα σε άλλους τομείς όπως η μουσική και τα βίντεο. Θα πρέπει να μην αναμειγνύουμε βέβαια τη συζήτηση του ΦΠΑ για τα βιβλία με την πρόταση την οποία έχουμε μπροστά μας και την οποία περιμένουμε για το τέλος του χρόνου. Συνεπώς λοιπόν και σχετικά με την δράση την οποία μας προτείνεται και σεβόμενη την αρχή της επικουρικότητας. Καμία χώρα δεν είναι υποχρεωμένη να το εφαρμόσει αυτό, αλλά έχει την δυνατότητα να προσαρμόσει τα επίπεδα ΦΠΑ αν το επιθυμεί και αν έχει μειωμένο ΦΠΑ για τα βιβλία. Ας προχωρήσουμε λοιπόν γρήγορα. Σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κάποιος από το ECR. η εκπρόσωπος των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Επιζητούμε ένα νομοθέτημα σχετικά και στέλνουμε πιστολές, πάρα πολύ εξήμων, πολύ άρα πάρα πολύ θετικό ότι υπάρχει αυτή η εύστοχη πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μα τι να πούμε στον κόσμο για τη διαφορά μεταξύ χαρτιού και ψηφιακών βιβλίων. Σύμφωνο. Πάντως με τον ε, εισηγητή να υπάρξει ταχεία εκεί πέρα στο Συμβούλιο και το θέμα να προχωρήσει. Ε, τον ευχαριστώ, τον εισηγητή. Μπράβο του για την έκθεσή του. Είναι πολύ σημαντικό το ότι αντιστάθηκε στον πειρασμό για όλες εκείνες τις τροπολογίες που δεν αφορούσαν ουσιαστικά το θέμα. Μπράβο που έμεινε στο κυρίως θέμα. Ελπίζουμε σύντομα να ολοκληρωθεί αυτή η διαδρομή. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε για την ε, Γκουε. Τώρα η Παλώμα Μπερμέχο δεν ήρθε, ούτε είναι κάποιος άλλος εδώ από την αριστερά. Πράσινη. Η κυρία Κέιτο. Όχι, σήμερα δεν θα διαφωνήσω γιατί συμφωνώ με όλα όσα προαναφέρθηκαν. Πολύ λογική η πρόταση. Συμφωνούμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά συμφωνούμε και με τις προσθήκες του εισηγητή. Το βιβλίο είναι βιβλίο και εφημερίδα εφημερίδα. Είτε είναι έντυπη, είτε είναι ψηφιακή. Τα κράτη-μέλη να έχουν ευελιξία για μειωμένο ΦΠΑ και για τα μεν και για τα δε. Και για τα ηλεκτρονικά βιβλία. Και αυτό νομίζω ότι μας βρίσκει σύμφωνος. Άρα νομίζω ότι αυτή η έκθεση θα προχώρησε χωρίς προβλήματα. Ήταν ενδιαφέρον το ότι μπορούσαμε να συνηθούμε με κάποιους εκδότες και να τα πούμε. Το πραγματικό πρόβλημα είναι η χρηματοδότηση των πολιτιστικών προϊόντων. Και είδαμε το ότι όντως χρειάζονται εφημερίδες υπήρξαν πολιτικά προβλήματα από το ότι το μοντέλο χρηματοδότηση δεν λειτουργήσε. Και συμφωνώ με την κόρα. Προσπαθήσαμε αυτό να το πέρασουμε στην έκθεση, αλλά τέλος πάντων να το δούμε στην Επιτροπή μας. Είδατε ποιο είναι το πρόβλημα των δημοσιογράφων. Δεν βγάζουν λεφτά εφημερίδε. Τι να κάνουν δημοσιογράφοι. Ε, εν τίποτα το με πτώγει αυτή την έκθεση. Συμφωνώ με τον εισηγητή. Ευχαριστούμε, λέει ο κύριο Φέρμπερ. Δεν βλέπω από το ΙΕΝΕΦ κάποιον, δεν βλέπω άλλον συνάδελφο που να ζητεί το λόγο. Όμω θέλει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Ραπόνια, θέλετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όχι, όχι, δεν έχω να προσθέσω τίποτε. Νομίζω ότι η θέση του Κοινοβουλίου είναι στο ίδιο μήκο σχήματο με τη δική μα πρόταση. Νομίζω το συντομότερο δυνατόν θα τα βρούμε στο Συμβούλιο. Ακόμα και αν αυτό δεν είναι αυτονόητο βέβαια τώρα που έχουμε τον κανόνα τη ομοφωνία. Ε, ευχαριστώ, ευχαριστούμε και εμεί, λέει ο κύριο Φέρμπερ. Κύριε Σιγητά, θέλετε κάτι. Κύριε Φάντε Ευχαριστώ να θυμάστε τη σημερινή μέρα. Είναι μοναδική πρωτοφανής περίπτωση ομόνιας και συνένεσης. Ε, για τα φορολογικά είναι ευκολότερο να βρούμε την ε, ομοφωνία εδώ παρά με το Συμβούλιο. Θα ψηφίσουμε στις 5 ώρα, 8 Μαΐου θα, το, θα ζητηθεί και, και θα κατέβει στην Ολομέλεια, δεύτερη Ολομέλεια του Μαΐου. Νομίζω ότι θα προχωρήσουμε συγχρονισμένοι με, με το ECOFIN. Πάμε τώρα στο σημείο 7 της μέσης της όσον αφορά αυτού του είδους τα υβριδικά μέσα με τρίτες χώρες. Όλε Λούντβιξον είναι ο εισηγητής, έχει το λόγο όλα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Για να μειώσουμε τη δυνότητα φορολογικού σχεδιασμού σε σημαντικό βαθμό, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ε, μια σειρά φορολογικών προτάσεων ώστε να φροντίσουμε οι πολυεθνικές εταιρείες με διασυνοριακή δραστηριότητα να πληρώνουν ε, τους φόρους που πρέπει εντός της Ευρώπης. Ε, οι βρυδικές ασυμφωνίες χρησιμοποιούνται συχνά για να ελαχιστοποιήσουμε την φορολόγηση των επιχειρήσεων και το είδαμε αυτό στην περίπτωση της Apple και το έχουμε δει και στην περίπτωση της McDonald's. Ε, τέτοιο είδος ερυθμίσεων χρησιμοποιείται με μοναδικό στόχο να ε, μειωθεί η φορολογία, κάτι που οδηγεί ε, σε υπονόμευση της φορολογικής βάσης των εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ε, αποτελεσματικοί κανόνες είναι απαραίτητοι λοιπόν ε, ώστε όσο μεγαλύτερος αριθμός ε, υβριδικών ρυθμίσεων να καλύπτεται από την νομοθεσία. Και γι' αυτό επικροτώ την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Συμφωνία του Συμβουλίου. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλύπτει τις ε, ασυμφωνίες ε, όσον αφορά την ε, φορολογική έδρα. Η περίπτωση της Apple δείχνει ότι είναι απαραίτητο να έχουμε πιο αυστηρούς κανόνες ώστε οι επιχειρήσεις να συμβάλλουν περισσότερο στο κοινό καλό. Ε, προτείνω η μόνιμη εγκατάσταση κατάσταση που δεν λαμβάνεται η υπόψη Ε, να μην λαμβάνεται υπόψη, διότι οι ασυμφωνίες μπορούν να οδηγήσουν σε διπλή έκπτωση ή έκπλωση χωρίς καταχώρηση και γι' αυτό δεν θα πρέπει να επιτρέπονται. Σε περίπτωση που η μόνιμη εγκατάσταση δεν λαμβάνεται υπόψη, θα πρέπει το κράτος μέλος, στο οποίο ο ε, πιστωτής έχει έδρα, να συμπεριλαμβάνει το εισόδημα το οποίο ε, κατά τα άλλα θα έπρεπε να αποδίδεται στην μόνιμη κατάσταση. Η περίπτωση της ε, McDonald's ε, δείχνει ότι δεν είναι αποδεκτή η κατάσταση. Οι συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας πρέπει να έχουν στόχο να οδηγήσουν στην αποφυγή της διπλής φορολογίας, όχι να έχουμε διπλή μη φορολόγηση. Σε θα πρέπει οι φορολογικές αρχέ να έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν σε περίπτωση που υπάρχουν φορολογικέ ασυμφωνίε και είμαι πεπισμένο ε, ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο να κλείσουμε τα παραθυράκια στα ε, ε, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ε, πρόταση της, του Συμβουλίου επιτρέπεται στα κράτη-μέλη ε, για περιορισμένο χρονικό διάστημα να ε, δώσουν παρέκκληση για τον τραπεζικό τομέα. Αυτό ε, Όμω ε, το κενό θα πρέπει να κλείσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του κοιόδε συζητητέ και τη γραμματεία τη ΕΚΟΝ για την καλή συνεργασία. Ελπίζω να μπορέσετε να υιοθετήσετε σήμερα τι ε, συμβαστικέ προτάσει μα ε, και να υιοθετηθούν στην Ολομέλεια το, στα τέλη Απριλίου. Thank you very much and... Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίνω τώρα το λόγο στους και οδησυγητές. Ελ Πιετικάινεν, παρακαλώ. Καταρχάς ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές ε, για την πολύ καλή συνεργασία. Η έκθεση αυτή νομίζω ότι ακολουθεί την διαγραμμή με την προηγούμενη. Εντός του Κοινοβουλίου λοιπόν δεν έχουμε σημαντικές διαφωνίες. Όλοι πιστεύουμε ότι η νομοθεσία θα πρέπει να καλύπτει τις ε, περιπτώσεις ασυμφωνίας, ε, δηλαδή τις ε, περιπτώσεις που, που αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μην έχουμε φοροαποφυγή. Νομίζω ότι έχουμε ελπίδες να πετύχουμε καλό και ισορροπημένο συμβιβασμό. Είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε την πρόταση. Ευχαριστώ. από το ECR, η Πύρκο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόταση οδηγίας για τις υβριδικές ασυμφωνίες είναι μια πρόταση την οποία επικροτούμε. είναι κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις τρίτες χώρες. Ευχαριστώ τον εισηγητή και, ο, και τους κοιόδης εισηγητές. Φαίνεται ότι όλοι έχουμε κοινό στόχο να εξαλείψουμε τις ε, δυνατότητες για φοροαποφυγή στην νομοθεσία μας. Πιστεύουμε Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους διάφορους ευρωβουλευτές σχετικά με το πώς θα το πετύχουμε αυτό. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να απαριθμίσουμε όλες τις πιθανές περιπτώσεις, ενώ κάποιοι άλλοι δεν πιστεύουμε ότι χρειάζεται να προβλέψουμε ήδη τώρα μελλοντικά παραθυράκια. Έχουμε όμως κοινό στόχο, γι' αυτό είμαι σίγουρη ότι θα βρούμε συμβιβασμό στην πρόταση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, από τους φιλελεύθερους, ο Νίλ Στόρβαλσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ και ο Λελούτβιξον για την πολύ καλή συνεργασία ήδη από την αρχή. Σε ευχαριστώ και για το καλό αποτέλεσμα. Φυσικά είναι πολύ τεχνικό το θέμα αυτό. Όπως γνωρίζουμε, ο διάβολος βρίσκεται στη λεπτομέρεια και στην περίπτωση αυτή. Είχαμε λοιπόν διάφορους διαβόλους. Προσπάθησα να υποβάλω κάποιες τροπολογίες ε, για να ενθαρρύνω τον Όλε να είναι πιο φιλόδοξος, ε, πιο τολμηρός. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω που έλαβε υπόψη του τις ε, τροπολογίες μου. Είμαι πολύ ικανοποιημένος ε, και νομίζω ότι έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να πω και πολλά άλλα. Είμαι ο πρώτος που θα υπερψηφίσω την έκλη αυτή και ελπίζω ότι καταφέραμε να βελτιώσουμε την νομοθεσία. Ελπίζω να έχουμε αποκλείσει κάποιες δυνατότητες φόρου αποφυγής Και αυτό είναι καλό. Άνοιξα σήμερα την έκθεση της Oxfam για να δω τι γίνεται στον τραπεζικό κόσμο και ο Όλε νομίζω ότι έχει ε, καταφέρει να δυσκολέψει κάπως τη ζωή των, ε, των επιχειρήσεων για φοροαποφυγή στο μέλλον. Ευχαριστώ, δεν βλέπω κανέναν από την ΚΟΕ. Την Ευαζολή αντικαθιστά η μόλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, μιλώ στο όνομα της Ευαζολή που επίσης ήθελα να ευχαριστήσει θερμά τον Όλε για τη δουλειά του πάνω στο ε, θέμα αυτό. Επίσης, ε, με χαρά διαπιστώνουμε ότι έχουν υιοθετηθεί οι τροπολογίες μας ε, και είμαστε ε, διατεθειμένοι να δεχτούμε όλους τους συμβιβασμού που προτείνει. Αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και βασίζεται στην οδηγία για την φοροαποφυγή που υιοθετήθηκε πέρσι. Ωστόσο, πρόκειται για μόλις ένα βήμα στο ταξίδι αυτό. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση για να Υιοθετηθούν ε, και άλλες προτάσεις, ε, όπως ε, για παράδειγμα τις συστάσεις αναχώρα, όπου έχουμε το, την φορολογία των επιχειρήσεων η Oxfam, υπολογίζει το πόσα χρήματα πηγαίνουν σε φορολογικούς παραδείσους από τις τράπεζες. Θα πρέπει λοιπόν οι προτάσεις μας να καλύψουν όλες τις επιχειρήσεις όσο γίνεται πιο γρήγορα. Πάντως είναι χρήσιμο να έχουμε αξιολόγηση τη συγκεκριμένη πρότασης μετά από τρία χρόνια από την ε, θέση σε ισχύ της, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι είναι αποτελεσματικά τα μέτρα αυτά και να ε, εντοπίσουμε ενδεχόμενα νέα παραθυράκια που θα έχουν δημιουργηθεί. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον εισήγητη και τους άλλους πιο για την πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτώ δεν ζητάει κανείς άλλο το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να πάρει το λόγο. Όλε. Για να κλείσεις ε, την ε, συζήτηση. Παρακαλώ. Ε, ναι, δεν θα μακρηγορήσω. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την ε, καλή συνεργασία που είχαμε με τους κοιόδης εισηγητές για το θέμα αυτό που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, ε, θα ήθελα να πω ότι στην νομοθεσία πρέπει πάντα να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Εγώ εργάστηκα σε μεγάλη επιχείρηση επί πολλά χρόνια και γνωρίζω ότι φυσικά προσπαθούν οι επιχειρήσεις ε, να ελαχιστοποιήσουν ε, τη φορολογία τους. Θα πρέπει λοιπόν συνεχώς να τροποποιούμε την νομοθεσία με βάση τα όσα συμβαίνουν στην πραγματικότητα στι διάφορες χώρες. Ε, Σα ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και πάλι όλους τους σκιώδεις συζητητές. Uh, Σε μισή ώρα θα γίνει η ψηφοφορία. Σε μισή ώρα, σήμερα. Και στη δεύτερη ολομέλεια του Απριλίου θα κατέβουν όλα Θα πάμε τώρα στο σημείο υπερθυμών. Αυτό λειτουργία δικαιόχρηση στον τομέα του λιανικού εμπορίου. Ο κύριο Ντόρ Κλόντιαν Φρουνσούλητσα είναι ο εισηγητής. Όμως δεν τον βλέπω στην έψο Ξέρει κάποιος άλλος από τους σοσιαλιστές. Ναι, ναι, ναι, Έρχεται, έρχεται. Βρίσκεται καθοδόν. Τι θα πει καθοδόν, θα πει να κάνουμε δίλεπτο διάλειμμα ή τι λέει ο κ. Πρόεδρος. να περιμένουμε τους σοσιαλιστές. Δίλεπτο διάλειμμα. We missed you. Please take a Το σημείο 8, η Ο κ. Φωνσουλίτσα είναι ο εισηγητής. Έχετε λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι. Να ευχαριστήσουμε πρώτα-πρώτα τους σκιώδες εισηγητές για την συνεργασία που ήταν πάρα πολύ καλή. δικαιώση είναι πολύ σημαντική για την ενιαία αγορά αλλά και για το λιανικό εμπόριο είναι πολύ σημαντικό θεσμό. Όμω δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τι δυνατότητε αυτού του θεσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω τη νομοθεσία που έχουμε. Δεν έχουμε εναρμονισμένη εφαρμογή του κανονισμού 330 του 10 δεν έχει αναρμονιστεί μεταξύ των κρατών μελών. Άρα δεν έχουμε αποτελεσματικότητα και νομίζω ότι έχουμε κάποιες συμβατικές προτάσεις. Σε αυτές καταλήξαμε σε συνεργασία με τους πιο ηγητές και καλύπτουμε έτσι τα πιο σημαντικά ζητήματα. Ε, λάβαμε υπόψη και όλες τις τροπολογίες και έτσι μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μια ενιαία αντιμετώπιση της δικαιόχρησης και ο κανονισμός 330 του 10 που σας προανέφερα θα πρέπει να εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κρατη Δεν έχουμε πληροφορίες για την εφαρμογή. Επομένως θα πρέπει τα κράτη-μέλη να φτιάξουν ένα μοντέλο υποβολής έκθεσης για καταγγελίες, για στοιχεία που έχουν αυτό μέσω κάποιων σημείων επαφής. Τέλος πάντων με οποιοδήποτε τρόπο. Έτσι να απλουστεύσουμε τη διαδικασία συλλογή πληροφοριών όσον αφορά το τι επικρατεί στην αγορά. Από την άλλη μεριά, συνάδελφοι, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει το να υπάρχει ισορροπημένη εκπροσώπηση των εμπλεκομένων στην δικαιόχρηση των δύο συμβολωμένων, ούτως ώστε να υπάρχει κάποιο είδου ε, ανεξάρτητη εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων όσον αφορά τις συμβάσεις δικαιόχρησης, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Προσφοράς. Και αυτό να αφορά και τον φορέα δικαιόγνωσης που υπάρχει σε επίπεδο ένωσης, αλλά και σε εθνικό επίπεδο επίσης. Θα πρέπει να διαμορφώσουμε πιο σωστά το νομοθετικό περιβάλλον των συμβάσεων. Να εξασφαλίσουμε την συμμόρφωση με την εργασιακή νομοθεσία, να υπάρχουν υπηρεσίες ποιοτικέ και αυτό με κατευθυντήριες γραμμές που θα αφορούν Τη Συμβάση Δικαιώσεω. συγκεκριμένα με του κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού από τα κράτη-μέλη. Ε, θα πρέπει αυτά να αξιολογηθούν και να θεωρηθούν. Επίση, να, γίνει μια αξιολόγηση του ποια είναι τα προβλήματα που προκύπτουν από τι νέε τάσει ιδίω όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ψηφιοποίηση. Επίση, σα τονίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει ενεργά να αναμειχθεί στην υπόθεση αυτή και στην περίπτωση που έχουμε οδηγίες και κανονισμούς για τη δικαιόχρηση και που έχουν προσαρμοστεί ούτως ώστε να υπάρχει ένα πιο λογικό, πιο αποδοτικό νομοθετικό πλαίσιο. Πάρα πολύ σημαντικό είναι και το εξής. Όσον αφορά το δίκαιο του ανταγωνισμού, θα πρέπει σε κάθε κράτο μέλο να κάτσουμε και να αναλύσουμε τι ισχύει. Και αυτό με έναν μηχανισμό αξιολόγησης μέσω των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού και έτσι να καταλήξουμε σε θεμητές ε, συνθήκες ανταγωνισμού. Αυτό θα πρέπει να επιβληθεί από τις αγορές μας. Σας ευχαριστώ και περιμένω πώς και πώς τα σχόλια σας. Στα γαλλικά συμπαθάτε με που άργησα, αλλά νόμιζα στις παραδέκα θα λάβω τον λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Φέρμπερ και τώρα το λόγο έχουν οι για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Λέει η κυρία Γκάλ Πέλτς. Ευχαριστούμε. Πολύ καλή δουλειά του κυρίου Φουντζούλικα. Και εδώ δεν είχαμε σημαντικά προβλήματα στη συζήτηση γιατί ως αφετηρία είχαμε ένα κοινό μήκος κύματος. Θέλαμε να αρθούν οι φραγμοί που εμποδίζουν το εμπόριο. Οπότε, οι τροπολογίες και οι συμβαστικές τροπολογίες προς τα εκεί κατατείνουν. Θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με τις συμβαστικές όχλησες, θα πρέπει να γίνουν κάποιες ε, τροποποίησεις στην νομοθεσία και θα πρέπει να υπάρχει ενοποιημένη, ενιαία μάλλον αντιμετώπιση επίσης. Θα πρέπει να δούμε και τα θέματα του δικαίου ανταγωνισμού όλο και περισσότερο οι εταιρείε εξαπλώνονται και πέραν των εθνικών συνόρων, άρα και θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι ενίος ο χώρος της εταιρικής δραστηριότητας, άρα θα πρέπει έτσι να προσαρμόσουμε και την νομοθεσία. Χρειάζεται μόνο προσαρμογή. Προσαρμογή δεν σημαίνει αναγκαστικά θέσπιση νέας νομοθεσίας. Απλώς θα πρέπει να βελτιώσουμε την λειτουργία των ισχυών των κανονισμών. Όπως είπε ο εισηγητής. Έχουμε το δίκαιο ανταγωνισμού. Έχουμε την πολιτική ανταγωνισμού της Ένωσης. Πολύ σημαντικά στοιχεία αυτά. Να δούμε τι τώρα θα ισχύσει σε αυτό το μέτωπο. Θα πρέπει να απαγορεύσουμε κάποιες ε, παράνομες δραστηριότητες. Να άρουμε τους φραγμούς που εμποδίζουν την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Άρα είναι πολύ σημαντική υπόθεση η εφαρμογή του κοινωτικού δικαίου από τα κράτη-μέλη. Προσοχή μόνο και στο χρονισμό, στο timing τέλο πάντων αυτών των αλλαγών. Ε, στην ΙΜΚΟ πάντως έγινε συζήτηση για παράνομες ε, πρακτικές. Έχουμε τροπολογίες σχετικά γιατί υπάρχουν παραθυράκια στην νομοθεσία. Αυτό το έχουν γνωρίσει κάποια κράτη-μέλη. Το πώς αυτές οι αθέμητες πρακτικές ε, είναι επιζήμιες. Οπότε έχουν ληφθεί κάποια μέτρα ή σχεδιάζονται μέτρα για την εμπλούση αυτού του προβλήματος. Πάντως τα μέτρα αυτά είναι διαφορετικά σε κάθε κρατός μέλος, οπότε και γι' αυτό θα πρέπει κάπως να βρούμε ε, κάποιο είδους ενιαίο πλαίσιο. Στο παρελθόν Είχαμε τέτοιε αθέμητες εμπορικές πρακτικές και όλοι ξέρουμε πόσο έχουμε τέτοια φαινόμενα πάρα πολύ διαδεδομένα τέτοιου είδους. Θα πρέπει επομένως τα κέντρα αποφάσεων να αναλάβουν δράση. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τη συνεργασία ναι, τους συναδέλφους, ε, έχουμε τις συμβατικές τροπολογίες. Τέλος πάντων αναμένουμε τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Όσακ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει ο κύριος Οζόγκ. Νομίζω ότι είναι μια καλή γνωμοδότηση η οποία υπογραμμίζει τα σημαντικά θέματα που έχουν σχέση με τα franchising. Ανάλυση των αγορών και ανάλυση των μακροπρόθεσμων πρόπτικων στην περίπτωση των προβλημάτων τα οποία μπορεί να έχουν οι εμπλεκόμενοι στην συναλλαγή, εμείς δεν θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις προτάσεις σαν πολωνική αντιπροσωπεία, γιατί πιστεύουμε ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι σε αντίθεση με τους νόμους επί του ανταγωνισμού. Δεν θα υποστηρίξουμε επίσης σαν Πολωνοί τις συμβιβαστικές G αγγλικό και O αγγλικό. δεν νομίζουμε ότι θα πρέπει να στηρίξουμε την πρόταση αυτή στο σύνολό της. Σας ευχαριστώ κύριε Όσοκ. Η Γκουε δεν είναι εδώ. Η πράσινη. Όχι, λέει η κυρία Σκοτ Κέιτο, δεν είμαι ενήμερη. <laughs> Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε το λόγο. Παρακαλώ να είστε σύντομος. Να επαναλάβουμε αυτά που είπαμε πριν, ότι τα προβλήματα του franchising δεν είναι θέμα ανταγωνισμού. Δεν είναι κυρίως θέμα ανταγωνισμού. Εμείς προσπαθούμε να δούμε τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόζονται οι κανόνες. Θα οργανώσουμε μία συνάντηση και μία μικρή διαβούλευση γύρω από αυτό. Να πω πάντως ότι το θέμα αφορά αν θέλετε εμπορικές πρακτικές ή πιθανώς τραυλές εμπορικές πρακτικές, αλλά δεν είναι κάτι που άπτεται του ανταγωνισμού άμεσα θα δώσω ξανά το λόγο στον κύριο Φραντζούλητσα. Να διαβεβαιώσω τους συναδέλφους ότι θα λάβω υπόψη μου τις θέσεις τους. Έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις μέχρι τώρα με τους κοιόδης και η θέση μας νομίζω είναι σαφής είναι μια καλή, αν θέλετε, ε, ένα καλό σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη της αγοράς του franchising στην Ευρώπη. Η ψηφοφορία στην ε, Κυρίαρχη Επιτροπή θα καθυστερήσει λίγο, αλλά εμείς θα ψηφίσουμε αμέσως. Δεν έχω κάτι εδώ για την ημερήσια διάταξη. 6 και 5 θα ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες, ε, μέχρι τότε θα διακόψουμε, αλλά δεν θα διακόψουμε γιατί θέλει η κυρία Μπερές το λόγο. Να κάνω ένα διπλό σχόλιο, να πω ότι ο εισηγητής των σοσιαλιστών ε, ήταν εγκαίρος εδώ, απλά είχαμε προχωρήσει πιο γρήγορα. Και για τον χρόνο ψηφοφορίας θα πρέπει να κάνουμε μία συζήτηση ξανά για το αν θα πρέπει να είναι τόσο αργά. Είχε αποφασιστεί από τους συντονιστές για να μπορέσουν όλα τα μέλη να είναι στις Βρυξέλλες, να γίνει μια τέτοια ψηφοφορία στις 6, αλλά μόνο την Δευτέρα. Καλό θα είναι να μην ψηφίζουμε καθόλου τη Δευτέρα βέβαια. Αυτό είπα. Βεβαίως αν έχεις παράπονα και αναφορές στη συνάντηση. Yeah. Okay. Ωραία λοιπόν. Ο ε, Γερμανός Πρόεδρος θα κάνει όλα στην ώρα τους.

Υπότιτλοι AUTHORWAVE Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Σας παρακαλώ να βάλετε την κάρτα σας ε, στη συσκευή και να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Still three colleagues to vote. Four colleagues to vote. Άλλοι τέσσερις συνάδελφοι παρακαλώ να ψηφίσουν. Ένας μας απομένει τώρα. Ωραία. Λήξη της ψηφοφορίας. Της δοκιμαστικής ψηφοφορίας. Λοιπόν, Θα ξεκινήσουμε να ψηφίσουμε πρώτα την δική μου έκθεση για το στατιστικό πρόγραμμα. Τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 6 υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση 6 της Επιτροπής Απασχόλησης, ΕΜΠΛ 6. Έναρξη ψηφοφορίας. Vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εγώ νομίζω ότι ήταν κατά το ΕΛ και συγγνώμη, δικό μου λάθος ήτανε. ΕΜΠΛ 7, υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση 7 τη επιτροπή Απασχοληση Έμπλεκτα έναξη ψηφοφορίας. Vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική DA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική M μη με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλ 12. Υπέρ. Γυρνάμε σελίδα. Υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Έμπλ 12. 12 τη επιτροπή Απασχόλησης Έναξης ψηφοφορία. Vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έμπλ 13 υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση 13 της Επιτροπής Απασχόλησης ενόψης της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΗ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική EA με προφορική τροπολογία. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν τη συμβιβαστική τροπολογία χωρίς την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 77 έχει αποσυρθεί. Συμβαστική L με προφορική τροπολογία. Πρώτα την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική L χωρίς την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προχωράμε στην τροπολογία Έμπλ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 25 υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση 25 της Επιτροπής Απασχόλησης. Έμπλη 25 έρχεται ψηφοφορία. Vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έμπλη 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση της τροπολογής 87 άρχεται η ψηφοφορία. Vote is Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Η 88 έχει αποσυρθεί. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική A, α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 2 υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση, η τροπολογία 2 της Επιτροπής Απασχόλησης. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά 33, η 33 καταπίπτει, 34 υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση της 34 έναξης ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έμπλ 3 υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση της τροπολογίας 3 της Επιτροπής Αποσχόλησης Άνξης Ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ή ε. Έχουμε πρώτα προφορική τροπολογία. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική χωρίς την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 4 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 20 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση της 20, έναξη ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία επάνω στο σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Έναρξη της ψηφοφορίας. Vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. 39 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, 4 αποχές. Ονομαστική ψηφοφορία πάνω στο νομοθετικό ψήφισμα. Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 43 υπέρ, μία κατά, δύο ε, αποχές και ψηφίζουμε την απόφαση να ε, ξεκινήσει διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο σύμφωνα με τον κανονα, ε, το, το άρθρο 1 γάμα του κανονισμού, έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 43 υπέρ, 0 κατά, 2 αποχές εγκρίνεται. Εγκρίθηκε η έκθεση, εγκρίθηκε και η, ε, η απόφαση να ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος σύντομα. Και τώρα πάμε στην έκθεση Λούντβιξον που αφορά τη μεταχείριση υβριδικών μέσων, της σχετικές ασυμφωνίες κατόπιν διαδικασίας ε, διαβούλευσης. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Για το 15 ψηφίζουμε. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10, 77 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Επαλήθευση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 Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για το 26. Ψηφίζουμε. Πέρασε φορείας. Εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική C. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Για το 86 ψηφίζουμε. Πέρασε. Όντω απορρίπτεται. 87 υπέρ, κατά. Έλεγχος για το 87. Πέρασε. Α, ισοψηφία Επομένω απορρίπτεται 31 και 32 υπέρ κατά αποχές συγκρίνονται, 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά εγκρίνεται 36 υπέρ κατά εγκρίνεται 37 υπέρ κατά έλεγχος για το 37 ψηφίζουμε πέρασε απορρίπτεται 38 υπέρ κατά Έλεγχος για το 37. Συγγνώμη, συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος, για το 38. Για το 38. Έλεγχος. Με ακούλπα, λέει ο Πρόεδρος. Ψηφίζουμε για το 38. Ηλεκτρονικά. Πέρασε. Εγκρίνεται. 39 συμβατή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 και 48 υπέρ κατά 49 υπέρ κατά το ΕΛΚ είναι κατά του 49 έλεγχος έλεγχος για το 49 πέρασε δεν 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Είστε υπέρ κατά του... Τέλος, θα κάνουμε έλεγχο για το 50. Σηκώστε το χέρι σας καθυστερημένα. I look at coordinator, but vote is closed. Πέρα ψηφοφορίας ε, και εγκρίνονται. Καλά που κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Μετά. 51 υπέρ. Υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβαστική ε υπέρ κατά ε, εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά. Έλεγχος για το 58. Σκώστε το χέρι σας παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Ήταν το 9 γιατί το 3 καταπίπτει 60 και 4 υπέρ κατά εγκρίνονται 61 και 5 και 62 όχι μόνο 61 και 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 62 υπέρ κατά έλεγχος για το 62 ψηφίζουμε Ε, απορρίπτεται, ναι. Απορρίπτεται και πάμε στο 63. 63 και η 6. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Πέρα Εγκρίνεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται, αλλά ας κάνουμε έλεγχο. Ψηφίζουμε. Και απορρίπτεται. Επτά υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Μάλλον απορρίπτεται. Ήταν οριακή η πλειοψηφία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Το 8 κατά 67 υπέρ, κατά, α, αποχές, α, απορρίπτεται. Συμβαστική F υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 71 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμφωνή, για το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε πέρασε 44-0 και με δύο αποχές συγχαρητήρια εισηγητά Και τώρα. Ψηφίζουμε το επόμενο. Yeah. We vote draft opinion by uh, Doru Claudian Frunzulitsan uh, Γνωμοδότηση Φρουντσούλητσα για τη λειτουργία δικαιόχρηστη franchising συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Παρακαλώ οι συντονιστές των δύο μεγαλύτερων ομάδων να συγκεντρωθούν λίγο. Συμβιβαστική B αγγλικό υπέρ κατά δεκτό. Τροπολογία 5 υπέρ <clears throat> κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 5 ψηφίζεται. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική C υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική ή υπέρ κατά αποχές δεκτή. 14 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 14. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική H υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική I υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική J υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική K υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική L υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική M υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική O υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ονομαστική κλίση τώρα. Στο κείμενο όπως τροπολογήθηκε ψηφίζεται. Τέλος της ψηφοφορίας. 42 υπέρ, ένας κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και τέλος, θα σας πω τι θα ψηφίσουμε. Τα πρίψ. για τις καταξιδότηση συμπράξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει ένα τίτλο πάρα πολλές σειρές, δεν θα τον διαβάσω. Υπάρχει μια πρόταση να ψηφιστούν όλα από κοινού. Εκτός από τις παραγράφους 1 και 2 και από το 1 μέχρι το H. Αλλιώς αν θέλετε ψηφίζουμε όλα αμπλοκ. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτά. Τώρα ονομαστική κλίση. One more to vote. If it's not mandatory. Okay, we close the vote. Τέλος της ψηφοφορίας. 41 υπέρ, 1 κατά μία αποχή. Οπότε η μία αντίρρηση γίνεται και αυτή δεκτή. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει την Δευτέρα 10 Απριλίου από τις 3 μέχρι τις 6.30 και 3η 11 Απριλίου από τις 9 μέχρι τις 12 και μισή. Σας ευχαριστώ όλους. Uh,